Guten Καλή μέρα, καλημέρα σε όλους. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μεγάλη αίθουσα και πολλοί απουσιάζουν δυστυχώς διότι ταυτόχρονα συμμετέχουν σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ψηφίζουν και τα λοιπά. Λοιπόν, δικαιολογούνται οι απόντες. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ αν είμαστε σε άλλη αίθουσα θα ήταν γεμάτη σίγουρα γιατί πολλοί βρίσκονται πίσω στις πίσω σειρές από τους ε, όσους συμμετέχουν. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έγκριση ημερησίας διάταξης πρώτα. Δεν υπάρχουν ενστάσεις, τώρα έγκριση πρακτικών. Εσείς κύριε Σάκε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Απλά και μόνο ήθελα μια προσθήκη στα πρακτικά να υπάρξει. Την τελευταία φορά όταν συζητήσαμε τη μειοψηφική άποψη δεν είχα την ευκαιρία να ανταποκριθώ και να τοποθετηθώ στα σχόλιά σας. Μια και βρίσκεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και θα έχουμε και πρακτικά, θέλω να διασφαλίσω ότι δεν θα υπάρχουν κάποιες ε, μη συνήθεις πτυχές όσον αφορά τους κανονισμούς και τις ε, Διαδικασίε Από πλευρά τη ομάδα μας είναι μειοψηφική η άποψή μας. Απόλυτα ομαλό και κανονικό αυτό. Εκπροσωπούμε τους εκπροσώπους μας σε εκλογικές μας περιφέρειες, σε ένα δημοκρατικό καθεστώς και είναι σημαντικό αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά. Έχετε δίκιο, λέει η Πρόεδρος. Πρέπει να πω και γι' αυτό κάτι κατά τα μέσα της ψήφισης, της ψηφοφορίας που δεν μπορεί να γίνει συζήτηση διαφορετικών απόψεων, στο τέλος είχατε ευκαιρία να το κάνετε όμως και εσείς και ο συνάδελφος ο δικό σα συνάδελφο τη Γκουε τη Ενωτική Αριστερά. Αλλά κανεί δεν ζήτησε να λάβει τον λόγο σηκώνοντα το χέρι του για την ψηφοφορία για να κάνει κάποια σχόλια. Εσεί πρέπει να ακολουθείτε του κανονισμού όπω και εγώ πρέπει να του εφαρμόζω. Την επόμενη φορά θα γνωρίζετε όταν θα υπάρχει ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία δεν μπορούν να συζητηθούν και να παρουσιαστούν διαφορετικέ απόψει. Μετά τι ψηφοφορίε μπορείτε να παρέμβετε εφόσον το επιθυμείτε για όσο διάστημα επιθυμείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ, λαμβάνετε υπόψη αυτό. Αν υπάρχουν κάποιες άλλες αντιρρήσεις σε σχέση με τα πρακτικά, μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης να μου το πείτε για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με την έγκριση των πρακτικών. Λοιπόν, επανέρχομαι στα γερμανικά και πάλι. Έχουμε διερμηνία, είναι εντάξει, φορέστε παρακαλώ τα ακουστικά σας, βάλτε τα ακουστικά σας. Thank you. Σήμερα έχουμε διαρμηνία. Δεν έχουμε, δεν έχουμε στα Ολλανδικά, ούτε στα Εσθονικά, Λιθουανικά, Λετωνικά, Μαλτέζικα και Σουηδικά. Δεν υπάρχει και διαρμηνία από και προς τα Κροατικά. Αλλά καταλαβαίνετε Γερμανικά εσείς, έτσι. Τέλεια, εξαιρετικά λοιπόν. Έχετε στους φακέλους σας, στα χαρτιά σας, μια σύντομη παρουσίαση για την τελευταία μας αποστολή Fact Finding Mission στην Φιλιππούπολη Πλόβδιβ στη Βουλγαρία από τις 9 11 Οκτωβρίου. Θα ήθελα να πω, δεν γνώριζα ούτε καν και το όνομα πιο πριν και ήμουν πολύ ε, ικανοποιημένη. Αν πάτε κάποτε στη Σόφια, βρεθείτε στη Μαύρη Θάλασσα, είτε από τη Μαύρη Θάλασσα επιστρέφοντας είτε από τη Σόφια. Αξίζει Φιλιππούπολη ένα ταξίδι. Είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει πολύ μεγάλη μακρά ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Χαίρομαι που πήγαμε στην Φιλιππούπολη και έτσι μπορούν αρκετά πράγματα να επεξηγηθούν για αυτή την Ευρώπη και για κάποιες γωνιές της Ευρώπης που δεν είναι τόσο γνωστές μας. Βλέπω στον κύριο Πιτέλα που είναι σπάνιος φιλοξενούμενος Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Θέλω να πω, έρχεστε εσείς από μια γωνιά της Ευρώπης που υπάρχει μια πολύ όμορφη πόλη που οι περισσότεροι δεν την έχουν γνωρίσει. Η Ματέρα, Ματέρα, όχι η Μαντέιρα, εντάξει. Ματέρα στην Μπαζιλικάτα, στην Απουλία, Πούλια. Πρέπει να ταξιδέψετε και να πάτε εκεί. Είναι μα την υποχρέωση. Στο μπάρι μπορείτε να πετάξετε στο μπάρι και από, με το αυτοκίνητο να πάτε στην ε, Ματέρα. Χαιρετίζω λοιπόν, αυτό ήταν σε σχέση με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, διότι και οι δύο, Φιλιππούπολη και Ματέρα, θέλουν να γίνουν πρωτεύουσες της Ευρώπης, πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Δεν πήγαμε όμως γι' αυτό εκεί, για να αναμειχθούμε σε αυτό, αλλά επειδή θέλαμε να γνωρίσουμε τη Φιλιππούπολη. Ξεκινάμε σήμερα με μια κρόαση που κανονικά πολλούς ε, θα ενδιαφέρει, δηλαδή ευκαιρίες, δυνατότητες ηλεκτρονικής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία, δημόσια κρόαση. Είμαστε για τις πολιτιστικές πτυχές εμείς αρμόδιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπως γνωρίζετε. Κυρίως είμαστε αρμόδιοι για την διάχυση και διεύρυνση και για τον πολιτισμό και την προστασία και αν θέλει κανείς να το πει έτσι για την προαγωγή των πολιτισμικών και πολιτιστικών πολυμορφιών της Ευρώπης και για την διασφάλιση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο στα κτίρια, αλλά και σε όλα όσα, όσα αφορούν την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών. Θέλω να υπογραμμίσω ότι έντονα ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Και όπως ξέρετε, η, εποχή της ψηφιακής, η ψηφιακή εποχή έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Και όλα αυτά χαρακτηρίζονται φυσικά από ταχύτατες εξελίξεις και μεταβολές και καινοτομίες από πλευράς τεχνολογίας που κάπως με κάνει να φοβάμαι και το λέω αυτό εξ αρχής ότι αυτό που όλοι πιστεύουν ότι όλα θα είναι ασφαλή όταν θα έχουν ψηφιοποιηθεί ίσως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι τόσο ασφαλή όλα αυτά διότι η τεχνολογία με άλματα, με αλματώδη πρόοδο ε, προοδεύει. Έχουμε σε αυτό το σώμα και την Ευρωπαϊκή που θα μεριμνήσει και θα φροντίσει η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να αποκτήσει ευδιάκριτο χαρακτήρα και να μπορέσει σε μία έδρα να παρουσιάζει αυτό το θέμα. Όταν έχουμε ένα πολιτιστικό, πολιτισμικό Google και που θα προαχθεί και θα διαχυθεί περαιτέρω και θα έχει ευρύτερο πλαίσιο από ένα Google, απλό Google, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ευρωπαίανα λοιπόν. Από ό,τι γνωρίζουμε όμως δεν είναι κάτι που από όλα τα κράτη να έχει επαρκώς ε, εξασφαλιστεί και ε, πρικοδοτηθεί. Είναι ακριβή αυτή η δαπανηρή διαδικασία. Δεν είμαστε εμείς που τα κάνουμε όλα. Οι χώρες πρέπει τα την ψηφιοποίηση να την προχωρήσουν και πολλοί διστάζουν ή δεν προχωρούν όπως πρέπει. Κάποιοι επέλεξαν το Google. Αν θυμάμαι καλά η Εθνική Βιβλιοθήκη στο Μόναχο ε, μέσα στο πλαίσιο της, του Google ε, ασχολήθηκε και όμως θέλουμε και εμείς να εμπλακούμε σε αυτό. Έχουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και ζητήματα ενώπιόν μας σε ένα κατάλογο. Προσκαλέσαμε επαΐοντες που θέλω να καλωσορίσω, τους χαιρετίζω. Ξεκινώ με τον κύριο δόκτορα Πέτερ Ντούσεκ, πρώην επικεφαλής από την Αυστρία ε, για τα αρχεία, τηλεοπτικά αρχεία και πρώην πρόεδρος της ΙΦΤΑ, Διεθνούς Ομοσπονδία Τηλεοπτικών Αρχείων. Μετά έχουμε τον κύριο Παλ Κέλλερ, αντιπρόεδρο της Knowledge Land από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Είναι μια ομάδα προβληματισμού, think tank, που σίγουρα προβληματίζεται για το ερώτημα, για το ζήτημα το οποίο σας παρουσίασα. Είναι όλα τόσο ασφαλή με την ψηφιοποίηση σήμερα ή όχι. Μετά με την Αν κυρία Αν Κατρίν Λογάν, που είναι ε, ερευνήτρια στο Ίδρυμα Max Planck για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για θέματα ανταγωνισμού όσον αφορά την ομοθεσία στο Μόναχο. Κάτι θα μπορέσει να μας πει για όλα αυτά τα θέματα. Μετά έχουμε τον κύριο δόκτωρα Στέφαν Γκράντμαν που είναι καθηγητής βιβλιοθηκονομίας και πληροφοριών βιβλιοθηκών όσον αφορά την Γερμανία στο Πανεπιστήμιο Humboldt Universität στο Βερολίνο σίγουρα όλοι είναι γερμανόφωνοι από ό,τι υποθέτω. Μπορούμε όμω και και να παρέμβουν στα αγγλικά. Στου φακέλους υπάρχουν κάποιε παρεμβάσει στα αγγλικά. Μπορείτε να παρέμβετε σε όποια γλώσσα επιθυμείτε. Αυτό καταδεικνύει ότι στον τομέα στον οποίο αναφέρθηκα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τέτοιε δράσει και θα πρέπει οι επαείοντε να συνεισφέρουν σε σχέση με αυτή τη δράση ευρωπαϊκή που είπα πιο πριν. Θα έχουμε την εξή διαμόρφωση την ακρόαση. Πρώτα, οι τέσσερι επαείοντε ανά τέσσερα λεπτά εκάστος θα μας εκθέσουν τις απόψεις τους. Μετά θα έχουμε μια ολόκληρη ώρα για ερωτήσεις, απαντήσεις από πλευράς μας. Και μετά θα έχουμε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να απαντήσουν οι πραγματογνώμονες σε παρεμβάσεις ε, και μετά θα έχουμε και εκπρόσωπο στο τέλος, ελπίζω τουλάχιστον από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου. Η Κύπρος θα ενδιαφέρεται φαντάζομαι ιδιαίτερα για αυτό το θέμα όσον αφορά και τα κτίρια Υπάρχει μεγάλος πλούτος σχετικά με την Κύπρο από πλευράς αυτής της πολιτιστική κληρονομιάς Και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται εξίσου και εδώ. Και ένα επιπλέον σημείο θα ήθελα να αναφέρω που όπως ε, αναφέρθηκε πιο πριν θα έχουμε την παρουσίαση στο διαδίκτυο της συνεδρίασής μας. Θα πρέπει λοιπόν σε σχέση με το μικρόφωνο που είναι αριστερά σας σε αυτό να στοχεύετε και να προσπαθείτε εκεί να ομιλείτε. Και όταν τερματίζετε την παρέμβασή σας να πατάτε το κουμπάκι, να σβήνει το μικρόφωνο σας ώστε ο επόμενος ομιλητής να μπορεί να παρέμβει και να ομιλήσει χωρίς πρόβλημα. Ξεκινάμε με τον δόκτωρα Πέτερ Ντούσεκ. Παρακαλώ έχετε τον λόγο κύριε Ντούσεκ. ich Μάλιστα. Μου ζητήθηκε να μιλήσω γερμανικά, έχω και στα αγγλικά το έγγραφο το οποίο κατέθεσα και πράγματι πολύ νωρίς άρχισα να ασχολούμαι με αυτά τα προβλήματα αυτού του θεματολογίου. Τυχαία, συγκυριακά, σε μια θέση βοηθού στο Βερολίνο, πέρασα στην παραδοσιακή, ας το πω έτσι, εκπαίδευση και κατάρτιση κατά την αρχή της δεκαετίας του 60. Και τότε ως αρχιονόμος μάθαινε κανείς τα μεσαιωνικά λατινικά για να μπορεί να τα διαβάζει και για την ε, ε, για τα χειρόγραφα ε, σε σχέση με την, ε, τις μεταγραφές με κεφαλαία ή και για τις φωτογραφίες που ξεκινούσαν τότε είχαμε χάσει 100 χρόνια των εξελίξεων. Είχαμε νέες πηγές που διασφαλίστηκαν αλλά δεν υπήρχε διαχείριση που να μπορούσε να είναι αποτελεσματική. Ήταν, ας το πω έτσι, τιμωρία κάποιος να πάει στα αρχεία αυτά και να δουλεύει εκεί. Ήταν, α το πω έτσι, δυσμενής μετάθεση. Ήταν εξορία εντός εισαγωγικών, ποινική εξορία. Χωρίς κονδύλια έπρεπε να εργάζονται με όλο και μεγαλύτερες στίβες και μεγάλες, ε, μεγάλα αποθέματα αρχείων. Είχαμε πολύ μικρά, μικρού εύρους ε, φιλμ, είχαμε βάρη μεγάλα τα οποία ε, συνεπαγόντουσαν όλα αυτά, ήταν κάτι για ασυβαρίστες όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά συνέβη, κάτι για την οπτικοακουστική κληρονομιά. Στην πρώτη φάση μόνο μπορεί κανείς ως πρωτομή να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια. Ε, όλοι φιλμάρισαν την ε, προσελήνωση στην σελήνη το 1969. Αλλά σε σχέση με τη δική μας δουλειά δεν γινόταν τίποτα. Υπήρχε, για, ας το πω έτσι, ε, η, προσελήνωση και όλα αυτά μας έθεσαν εμάς, μας, μας επισκίασαν. Πουθενά λοιπόν δεν είχαν όλα αυτά ε, από πλευράς μας ε, για τη δουλειά μας αποθηκευτεί. Βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή και τώρα υπήρχαν αυτοί οι φτωχοδιάβολοι που είχαν τα προβλήματά τους και που κανείς δεν τους έδινε κονδύλια και κανείς δεν μπορούσε να τους δώσει ένα πρόγραμμα να κάνουν κάτι αποτελεσματικό και κανείς δεν ενδιαφερόταν να μάθει τι γινόταν με αυτά τα αρχεία. Υπήρχαν τεράστια κενά. Μετά ήρθε ο κύριος Ντούσεκ που δεν πήγε ε, στο Βερολίνο αλλά εκπαιδεύτηκε ως αρχαιονόμος και ξεκίνησε με αυτή την εκπαίδευση και κατά τη διάρκεια των μέσων της δεκαετίας ε, ε, των 70 ξεκίνησε να εργάζεται μέσα στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης. με την ε, ενασχόλησή του με αυτά τα αρχεία με έναν πίνακα επιθυμιών και έργων που έπρεπε να επιτευχθεί υπήρχε και ένα μεγάλο κουτί το οποίο θα μπορούσε να τα εμπεριχεί όλα αυτά και μετά είδαμε ότι σε σχέση με όλα όσα ζητούντο δεν ήταν διαθέσιμα. Απλά πράγματα όπως γεωργοί για παράδειγμα που όργωναν με λογά τους ε, και μετά εδώ υπήρξε μία ας το πω έτσι τομή και προσπάθησα όλα αυτά να μπορέσουμε να τα θέσουμε σε τάξη συμβολικά ας το πω έτσι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η αρχή ήταν για μένα πραγματικά ένα πλήγμα στο τέλος τέλος όμως είχαμε ολόκληρες βαλίτσες από υλικό για την, τα μαθήματα ιστορίας ε, στα σχολεία. Και η πρώτη λέξη ήταν προστασία δικαιωμάτων δημιουργού και συγγραφέα. Και αν κάποιος ήθελε τα ε, δευτερογενή δικαιώματα για την προστασία όλων αυτών των προϊόντων όσα, όσον αφορά την ψηφιοποίηση ακόμα δεν γινόταν λόγος για ψηφιοποίηση ήταν ας το πω έτσι επιτυχία αν καταφέραμε να, να ξεπεράσουμε τα πρώτα προβλήματα. Ήταν όμως τόσο θελκτικά όλα αυτά που οι αυστριακοί ε, δάσκαλοι μπόρεσαν να ενασχοληθούν με αυτά για την ιστορία με ταινίες, ε, με διαγράμματα, με υλικό το οποίο ήταν πολύ καινούριο για μας. Και από όλα αυτά είχαμε μία σειρά web επταετούς διάρκειας ε, για την κάλυψη του κενού, του κενού στο ιστορικό αρχείο και τη διασφάλιση της ε, οπτικοακουστικής ε, ιστορικής κληρονομιάς. Προσπαθήσαμε αυτή την κατάσταση που έπρεπε να τερματιστεί, που δεν είχαμε ειδικού να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Και αυτό τι ήταν. Αν δει κανεί τι συνέβη από το 82 στο 88 ήταν μια τομή. Το 89 έγινα επικεφαλής ε, των, ε, τηλεοπτική, τηλεοπτικής υπηρεσίας με τελείως νέες ε, δομές και δυνατότητες. Και στο τέλος το επιστέγασμα ήταν το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Το 91 μια πολύ νεότερη ιστορία σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε ή προβλέπαμε. Όλα αυτά άμεσα βραχυπρόθεσμα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση, ιστορική κατάρρευση ενός ολόκληρου καθεστώτος. Πιστεύαμε ότι δεν θα υπήρχαν πλέον προβλήματα, ότι όλα τα προβλήματα θα είχαν επιληθεί, δεν θα υπήρχαν προβλήματα στο μέλλον και θα πνιγόμαστε στην εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση και πολιτισμό. Και πολύ γρήγορα προσγειωθήκαμε ότι δεν συνέβαινε αυτό πραγματικά. Προϋπόθεση όμως ήταν να έχουμε και τις δράσεις μας ε, ώστε νομοθέτες, νομο, πραγματογνώμονες ε, νομικοί να μπορέσουν να παρέμουν για τη διασφάλιση αυτών των αρχείων. Οι νομικοί εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Οι μεν είναι εκείνοι που προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο από μια περίπλοκη και δύσκολο να αντιπαρατεθούμε με αυτήν την κατάσταση και οι άλλοι βρίσκονται στην άλλη πλευρά και βοηθούν με προτάσεις ε, να προχωρήσουμε ώστε να μην συμβεί εκείνο το οποίο, ε, ε, στο οποίο στοχεύουν άλλοι. Ε, βλέπουμε λοιπόν τη διαφορετική λοιπόν προσέγγιση για το τι πρέπει να προστατευτεί και πώς πρέπει να προστατευτεί. Πολύ γοργά μπόρεσα να εμβαθύνω σε σχέση με, αυτές τις, ε, με αυτούς τους προβληματισμούς. Η Ολλανδία το έχει πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη αυτό όταν ξεκινήσαμε και πάλι η Ένωση ήταν ένα σύλλογος ή μια ένωση ε, συνταξιούχων αρχιοθετών που ε, είδαν το τι πρέπει να γίνει δεν είχαν ούτε καν ε, ένα ε, βίντεο, δεν είχαν κάμερα για να βιντεοσκοπήσουν, δεν υπήρχε εξοπλισμός. Είχαν ενασχόληση με εκπομπές στην τηλεόραση για την παιδεία και εκπαίδευση και κατάρτιση. Όλα αυτά μας ανάγκασαν τη δική μας ένωση να την θεωρούμε μια ένωση για ε, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση με δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ε, βιντεοσκοπημένες εκπομπές, ε, να χρησιμοποιούμε ψηφιοποιημένες εκπομπές και όλα αυτά βρίσκονται πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Τα CDs μπορεί να πει κανείς ότι όταν η ποιότητά τους μετά από πολλά χρόνια χρήσης ε, υποβαθμίζεται. Με την ψηφιοποίηση πρέπει λοιπόν να αντικατασταθούν γιατί δεν μπορούν να παίζονται πια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και φαίνεται ότι βραχυπρόθεσμα μπορεί να διασφαλιστεί αυτό. Για τις τεχνικές διαφορές ε, σε σχέση με τα προβλήματα των μηχανών και του εξοπλισμού που αναπαράγουν αυτές τις ε, εκπομπές. Πού βρισκόμαστε τώρα. Όλοι επιθυμούσαν να έχουμε σύγχρονα μέσα. Στη δεκαετία του 90 ως ε, σύλλογος, ως ένωση, είχαμε μεγάλες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Έπρεπε να αναζητηθούν κονδύλια και μέσω εξορθολογισμού και δράσεων εξορθολογισμού προσπαθούσαμε να τα διασφαλίσουμε και μετάθεση έργου. Και στην Αλβανία π.χ. παντού είχαμε, ας το πω έτσι, την, τα ε, σύγχρονα αρχεία τηλεοπτικών μέσων. Όλα αυτά τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι οι διαφορές οι πολιτισμικές ε, της Ευρώπης, η Ευρώπη των περιφερειών, χωρίς τα οπτικοακουστικά δεν μπορεί ούτε να διασφαλιστεί αυτή η κληρονομιά, ούτε να διατίθεται ε, στους πολίτες. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ψηφιοποίηση. Χρειαζόμαστε όλους για τους εξής λόγους κοινέ λύσεις. Δεν είναι δυνατόν οι επιτυχίες της Google χωρίς οποιαδήποτε προστασία ε, πνευματικών ε, δικαιωμάτων να προάγεται με αυτούς τους ρυθμούς. Δεύτερον, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις επιμέρους χώρες για τη δημόσια πρόσβαση και προσπελασιμότητα μιας χώρας σε αυτά, σε αυτά τα κομβικά σημεία. Για παράδειγμα, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της ε, Γαλλίας, για παράδειγμα, με την μεταφορά ε, προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων στα αρχεία, μετά από μια σειρά ετών ε, χάνονται αυτά τα πνευματικά δικαιώματα, παραγράφονται πλέον. Θα πρέπει έτσι λοιπόν να δούμε ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μη διαθέσιμων αρχείων και διαθέσιμων αρχείων με προσπελασιμότητα για το κοινό. Τεράστια διαφορά από χώρα σε χώρα και σε σχέση με την προσπελασιμότητα που πολλές φορές ε, ε, είχαν ε, εθνικοποιηθεί εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, τα δικαιώματα αυτά με την ψηφιοποίησή τους. Η κραυγή λοιπόν, η απέτηση να υπάρξει μια κοινή στέγη και ένα κοινό πλαίσιο στην Ευρώπη για την προστασία αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων και στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι σημαντική υπόθεση διότι στη συνεδρίαση για τα πνευματικά δικαιώματα με την ψηφιακή αυτοματοποίηση μάθαμε ότι για τα πνευματικά δικαιώματα κανείς δεν είναι τελικά ο μόνος αρμόδιος είναι η υπεύθυνοι για τα πολιτισμικά, πολιτιστικά θέματα ή ποιοι είναι. Είναι μια μεθοριακή, συνοριακή περιοχή μεταξύ ιδιωτικού δικαίου και δικαιωμάτων και δικαιωμάτων για την παιδεία και εκπαίδευση. Και τώρα έχουμε μία λύση για τη, τη βιβλιοθήκη, για το Ίδρυμα Σύγχρονης Ιστορίας, που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι φοιτητές στα αρχεία ψηφιοποιημένες λύσεις, αλλά μόνο για υλικό το οποίο έχει αποσταλεί σε εμά. Αυτό είναι σημαντικό για την χρήση των, ε, του υλικού που ε, εκπέμπεται. Ποτέ τα βασικά, τα, ε, όλα τα στοιχεία που έχουμε δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε άμεσα και ταυτόχρονα. Θα πρέπει να προστατεύεται η προστασία του απορρίτου. Και χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή λύση που θα ισχύει σε σχέση με τις ε, εκπομπές, το εκπαιμπόμενο υλικό, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σήμερα και για τις εφημερίδες και τα άρθρα τους. Δεν είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά είναι περίπλοκο στην υλοποίηση. Δεύτερον, όσον αφορά με ένα κατάλογο, να βλέπει κανείς πού υπάρχει τι, που θα πρέπει δωρεάν στο διαδίκτυο να είναι διαθέσιμο, όπως οι κατάλογοι βιβλιοθηκών. Αν ελεύθερα θα μπορεί κανείς να επιλέγει και να ε, έχει πρόσβαση στο πλήρες ε, περιεχόμενο όλων αυτών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε πώς θα γίνει. Ένα, ένα είναι σαφές. Όταν θα έχουμε μεγάλες όπερες, ε, τραγούδια, γνωστές παραγωγές που θα μπορούν ε, χωρίς ε, αμοιβή, χωρίς αντίτιμο να ε, είναι σε ελεύθερη πρόσβαση. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν αυτά. Έχουμε ένα κομβικό σημείο εδώ το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει εκ βάθρων και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Ευγνώμονες θα είμαστε αν μπορούσε αυτό να γίνει με πολύπλευρη συμμετοχή. Τώρα για την απέτηση να μπορεί κανείς όταν τρία σέντ εμβάζει κάποιος σε κάποιον άλλο ή σε σχέση με μια τέτοια συναλλαγή έχουμε 5 cents όλα όλα δεν είναι επαρκή δεν, ποσά, δεν από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με την αύξηση ενός τον καθορισμό ενός καταποκοπήν ποσού και όταν έχουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία και αυτό μας δίνει μια ιδέα το πόσοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αντλούν από τα αρχεία αυτά τέτοια, τέτοιο υλικό, όταν φτάσουμε σε τέτοια ρύθμιση, εγώ είμαι υπέρ της ρύθμισης με προσκαλέσατε, έχω προσκληθεί για το έτος ε, Verdi Wagner να ε, μπορέσω να δω τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τα αρχεία. Και εγώ 68 ετών ως συμμετέχον σε αυτό το κίνημα πρέπει να πω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι ένα είδος quiz που πρέπει να γίνεται δημόσια. Οι νεότεροι συνάδελφοι οι οποίοι ε, είχαν ε, ε, εμπλακεί. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιήθηκαν. Πρέπει κανείς παίζοντας σαν ένα παιχνίδι να μπορεί να ενασχολείται με αυτά. Ας μην ψάχνουμε να βρούμε μια τελεσίδικη συνολική λύση για όλες τις χώρες που θα ρυθμίζει τα πάντα. Ας μεριμνήσουμε για το έτος Βέρντι Βάγνερ ή ας ασχοληθούμε με το, το Ίδρυμα της Ιστορίας, σύγχρονης ιστορίας για να έχουμε μια κλιμακωτή, κλιμακούμενη, διαβαθμιζόμενη πρόσβαση να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες βήμα προς βήμα και να λιάνουμε το έδαφος. Πιστέψε με, δεν θα χρειαστούν άλλα 30 χρόνια για να επιληθούν αυτά. Πιέζει ο χρόνος, είναι αφάνταστη η πίεση ώστε να ξεπεράσουμε αυτά τα ψηφιακά εμπόδια και να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ήταν μια επισκόπηση ιστορική των πραγμάτων αυτή και ε, έχω την ηλικία να πω ότι τα έζησα, τα βίωσα όλα αυτά. Και είναι πράγματα τα οποία πριν από 15 χρόνια δεν θα μπορούσε να τα έχει φανταστεί κανεί. Πρέπει να πορευτούμε, να οδεύουμε με τις εξελίξεις, με την ε, χρονική συγκυρία στην οποία ζούμε ιστορικά και θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια δυνατότητα ευρωπαϊκά να δράσουμε αποτελεσματικά. Ξέρετε όμως ότι είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου αυτό διότι και στη μουσική και στις ταινίες και στα ντοκιμαντέρ πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν μπορεί αυτό γραμμικά να γίνει. Πρέπει πολύ πιο διαφοροποιημένα να εργαστούμε με μεγάλη φροντίδα και προσοχή ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες διαφοροποίησεις. Και με τις μικρές ή τα μικρά ατομικά αιτήματα διαδραματίζουν και αυτά ένα σημαντικό ρόλο. Έχουμε και ένα συνολικότερο πλαίσιο που έχει το βάρος του. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Δύο παρατηρήσεις. Μπορείτε να ακούσετε κροατικά, αγαπητέ συνάδελφε Μάτισεκ, και εσείς μπορείτε να μιλήσετε Ολλανδικά. Γίνεται αυτό λοιπόν. Πολύ ωραία. Ο κύριο Κέλλερ έφυγε. Α, όχι, εκεί πίσω είναι. Πολύ καλά. Κύριε Κέλλερ, εσεί είσαστε ο αντιπρόεδρο τη Knowledge Land της, χω... χώρας για τη γνώ... της γνώσης στο Άμστερνταμ. Έχετε τον λόγο για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Um, thank you very much for the... Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετοίμασα εισήγηση η οποία εδράζεται την εμπλοκή μας σε σχέδιο ψηφιοποίησης στις κατοχώρες, όπως είπε ο συναδελφός μου από το 2005, πάνω σε ένα μεγάλο έργο ψηφιοποίησης, το Images for the Future, εικόνες για το μέλλον, που αξιοποιεί υλικό από μουσεία, βάσεις δεδομένων, τα εθνικά αρχεία, φωτογραφίες μεταξύ άλλων και επιπλέον η Κένισλαντ τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή κυρίως πάνω σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, προστασίας τους και βεβαίως στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος προστασίας της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχω ετοιμάσει και ένα PowerPoint, ελπίζω να φαίνεται. Έχω προσθέσει και μια διαφάνεια για να αποτυπώσει το πρόβλημα καταρχήν. Την δείξαμε πριν δύο εβδομάδες σε μια άλλη διάσκεψη και παντά στο αν είναι διαθέσιμα τα αρχεία στο κοινό. Η απάντηση είναι όχι ακόμη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 97.000 περίπου, αν θέλετε, ώρες ταινιών και βίντεο αυτή τη στιγμή μόνο 17.300 ώρες είναι διαθέσιμες στην εκπαίδευση, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία μπορούν φυσικά να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο σκοπός είναι το υλικό αυτό, όλο το υλικό αυτό, να είναι διαθέσιμο. Ήδη 859 ώρες έχουν ψηφιοποιηθεί και θα μπορούσαν με ένα κλικ να διατηθούν στο διαδίκτυο. Θα τις βρείτε προς το παρόν στο euscreen.eu ή στο openimages.eu, μια Ολλανδική πλατφόρμα και φυσικά στο YouTube. Αυτό καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, πόσο περιορισμένες είναι οι τεχνικές μας δυνατότητες, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με το διαθέσιμο υλικό. Επιστρέφω όμως σε αυτό που θέλω να πω στην αρχή. Θα σας πω καταρχήν λίγα πράγματα για την πόλη μου, το Άμστερνταμ. Αυτό που βλέπετε είναι αεροφωτογραφία του Museum Plain, της πλατείας του Μουσείου στο Άμστερνταμ. Εκεί γύρω βρίσκονται τα διασημότερα μουσεία, όπως το Van Gogh, το βλέπετε εδώ, το Κρατικό Μουσείο, το Δημοτικό Μουσείο, εδώ, το οποίο φιλοξενεί συλλογές σύγχρονη και κλασικής τέχνης και το Rex Museum, το οποίο είναι το Εθνικό Μουσείο των Κάτω Χωρών που φιλοξενεί κατά κύριο λόγο συλλογές 17ου αιώνα της χρυσή εποχής της τέχνης στην περιοχή. Αυτό το οποίο ίσως δεν βλέπετε τόσο εύκολα βλέπετε εδώ τα δύο μάλλον και τα τρία μουσεία εδώ εδώ έχουν συγκεντρωθεί στον ίδιο χώρο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ένα τέτοιο μουσείο κλείσει για 10 χρόνια λόγω επισκευών. Η συλλογή θα μπορούσε να διατίθεται επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα δύο μουσεία από τα τρία δημιούργησαν ιστοσελίδες για την περίπτωση ακριβώ ε, έργων, για παράδειγμα, για την περίπτωση που είναι κλειστά, ώστε να μπορούν οι επισκέπτε να τα επισκέπτονται επιγραμμικά. Και αν ε, έρθουμε λίγο πιο κοντά στο Rex Museum, συλλογέ του 17ου αιώνα όπως είπα, ε, το μουσείο αυτό την περασμένη εβδομάδα άνοιξε την καινούργια του ιστοσελίδα, μια συγκλονιστική ιστοσελίδα, έτσι θα έπρεπε να είναι όλες οι ιστοσελίδες, όλοι οι ιστότοποι πολιτισμικών ιδρυμάτων, ρίξτε μια ματιά. Εάν κάνετε κλικ πάνω σε ένα έργο, θα το δείτε στο κέντρο της οθόνης. Υπάρχουν χιλιάδες ε, αναπαραγωγές υψηλής, σε υψηλή ανάλυση που θα απολαύσετε ανεξαρτήτως της ανάλυσης και του μεγέθους της οθόνης σας. Μπορείτε να κάνετε zoom σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, σε οποιοδήποτε βάθος, σε οποιαδήποτε ανάλυση και υπάρχουν εργαλεία για να αποκόψετε ένα τμήμα αυτού που βλέπετε στην οθόνη, να το χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες, μπορείτε να τυπώσετε, μπορείτε να τυπώσετε πάνω σε ε, φλιτζάνια, σε άλλα αντικείμενα, οπουδήποτε. Ο ιστόρροπος σας ενθαρρύνει, με άλλα λόγια, με δεκάδες τρόπους να επισκεφθείτε τον ιστόρροπο του μουσείου, να τον περιδιαβείτε, είναι ένα ιστότοπο ο οποίο ε, χρησιμοποιεί στο έπακρο όλε τι τεχνικέ δυνατότητε που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα. Θα δείτε επίση ότι το περισσότερο υλικό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ανήκει στην δημόσια σφαίρα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον πνευματικά δικαιώματα. Το μουσείο δεν δεσμεύεται από κανέναν περιορισμό περί πνευματικών δικαιωμάτων. Συγχαρητήρια στο Ρίξ Museum. Διότι από εδώ και πέρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με το υλικό ακριβώς επειδή δεν υπάρχει copyright, δεν υπάρχει προστασία. Έτσι όμως επιτελούν, εκπληρώνουν τη δημόσια αποστολή τους που είναι να δώσουμε στο κοινό όσο περισσότερα μπορούμε. Σε καιρό οικονομικής κρίσης και συρρυκνούμενων προϋπολογισμών σε καιρούς ε, όπου όλοι προσπαθούν να αυξήσουν τα κέρδη τους, τα έσοδά τους από τις συλλογές τους, αυτό αποτελεί ένα διαφορετικό παράδειγμα. Το μουσείο έκρινε όμως ότι μπορεί να έχει ένα μικρό σχετικά έσοδο από τις επαγγελματικέ χρήσεις, Σε αυτήν την περίπτωση το υλικό χορηγείται σε πάρα πολύ ψηλέ αναλύσει, αλλά αυτό είναι για του επαγγελματίε. Το υλικό υπάρχει σε υψηλή ανάλυση για όλους όμως εδώ και πολύ καιρό πριν καν εκπνεύσουν τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι ένας ιστότοπος του συγκεκριμένου μουσείου που δημιουργήθηκε για να δείξει την συλλογή του όταν είναι κλειστό. Το μουσείο θα ξανανοίξει 13 Απριλίου του 2013. Το κτίριο είναι συγκλονιστικό. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να το επισκεφτείτε. Ε, μην επισκεφτείτε μόνο τον ε, ιστότοπο. Πάμε τώρα στο Δημοτικό Μουσείο. Η εικόνα αυτή του Google είναι κάπως ε, ξεπερασμένη. Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Το μουσείο είναι ανοιχτό εδώ και ένα μισή μήνα με μεγάλη επιτυχία. Άρα μπορείτε να επισκεφτείτε τη συλλογή στο φυσικό της χώρο. Και το μουσείο αυτό όμως δεν ήταν προσπελάσιμο για πολύ καιρό. Προσπάθησαν λοιπόν να διαθέσουν την συλλογή τους στο διαδίκτυο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ειδού το αποτέλεσμα, ειδού αυτό που θα δείτε στον ιστότοπο του μουσείου, κάνετε κλικ στην επιγραμμική συλλογή. Θα δείτε μάλιστα τα γκρίζα τετράγωνα, τα οποία λένε ότι οι συγκεκριμένοι πίνακες δεν είναι διαθέσιμοι λόγω προστατευμένων πνευματικών δικαιωμάτων. Εδώ βλέπετε τα σύμβολα τα οποία σας ε, καθοδηγούν για να κάνετε zoom στη συγκεκριμένη εικόνα. Υπάρχει μια συλλογή 20ου αιώνα. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού στο Δημοτικό Μουσείο προστατεύεται από copyright για αυτούς είναι πολύ δύσκολο να έρθουν σε επαφή με τους ε, κατόχους των δικαιωμάτων για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το οποίο θα ήθελαν να κάνουν για το κοινό ή τους ε, ειδικού, ώστε να περάσουν πρόσβαση δηλαδή στο υλικό. Προσπαθούν σκληρά, πολλές φορές όμως ε, όπως στην περίπτωση αυτή Μπορεί κανείς να επισκεφτεί το έργο και να το δει στο φυσικό του χώρο, όχι όμως επιγραμμικά. Το μόνο που βλέπετε δηλαδή στον ιστόρπο είναι αυτό. Και αυτό λόγω της διαχείρισης των ε, δικαιωμάτων είναι αυτό το οποίο προανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Οι διαχειριστές των δικαιωμάτων στο παρελθόν δεν είχαν στο μυαλό τους το επιγραμμικό περιβάλλον, το διαδίκτυο δεν σκέφτηκαν, τώρα που δεν υπήρχε διαδίκτυο, να αγοράσουν μαζί με το έργο και τα επιγραμμικά δικαιώματα. Έτσι, δύο συλλογέ μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική τύχη, τελείως διαφορετική προβολή. Προσπαθήσαμε κάπως όλα αυτά να τα οργανώσουμε και εδώ η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Αν δούμε τις συλλογές των μουσείων, θα τις χωρίζαμε ως προς τα χαρακτηριστικά τους στα λεγόμενα μεταδεδομένα που εν γέννη καλύπτονται από το copyright του μουσείου για παράδειγμα από εκεί πέρα όσον αφορά τα δικαιώματα έχουμε τα αντικείμενα δημόσια όπως το Museum σε άλλες περιπτώσεις το copyright τα δικαιώματα ανήκουν στο μουσείο και στην τρίτη περίπτωση τα δικαιώματα, όπω γίνεται στι περισσότερε περιπτώσει, ανήκουν σε κάποιον τρίτο. Για τα έργα στη δημόσια σφαίρα και για την Ευρωπαία ναι, προκειμένου δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ίδιο ίσω ισχύει και με τι περιπτώσει όπου το μουσείο είναι κάτοχο των δικαιωμάτων. Το μουσείο αποφασίζει τι θα διαθέσει στο διαδίκτυο ή αλλού. Όλα αυτά καλύπτονται από την οδηγία περί ενημέρωσης του κοινού, μόνο που εκεί πρέπει να συμπεριλάβουμε και την πολιτιστική κληρονομιά στο πεδίο της εφαρμογής. Ξέρω ότι υπάρχουν σημαντικές αντιστάσεις εμπροκειμένου από μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, όμως μακροπρόθεσμα αν δούμε τα πλεονεκτήματα πιστεύω ότι από εδώ έχουμε να κερδίσουμε όλοι. Είναι σίγουρο ότι πρέπει και αυτό τα μουσεία, για παράδειγμα, να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ένα δημόσιο ρόλο, μια δημόσια εντολή αν θέλετε, που σημαίνει ότι η αποστολή τους είναι να διαθέτουν το υλικό αυτό στο κοινό. Το κοινό να έχει πρόσβαση και βεβαίως κάποιοι άλλοι να κάνουν σπουδαία δουλειά πάνω σε αυτές τις συλλογές. Τι γίνεται όμως με τα έργα των οποίων τα δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους. Δεν είναι κάτι που συζητούμε βεβαίω αυτή τη στιγμή, ούτε υπάρχει σχετική συζήτηση στην Κομισιόν. Η σχετική οδηγία καλύπτει ένα μικρό μέρο μόνο αυτών των δικαιωμάτων, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση όχι τα πάντα. Αν δούμε την ε, Ευρωπαϊκή, δείτε την κατανομή, είναι ο αριθμό των αντικειμένων κατανημένων ανά αιώνα. Και βλέπετε ότι τα περισσότερα αντικείμενα της συλλογής ανήκουν στον 20ο αιώνα, επειδή, έχει επειδή έχουν εκπνεύσει τα δικαιώματα. Στον 20ο αιώνα, από πλευρά δικαιωμάτων, πάρα πολλά έργα δεν την χάνουν προβολή ακριβώ λόγω δικαιωμάτων. Και το συμπέρασμά μου, εμπροκειμένο, για αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι ότι η μόνη πραγματική λύση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα είναι να προβλέψουμε εξαίρεση για τα πνευματικά πολιτικά ιδρύματα ώστε να μπορούν να προβάλλουν τα έργα τους για μη εμπορικούς σκοπούς επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Ιστορικός κάθε φορά που είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ προστασίας των δικαιωμάτων και ενό κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης προβλέψαμε απλούστερα εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις για αυτές τις χρήσεις, τις άλλες χρήσεις αν θέλετε. Η εκπαίδευση, ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένας τέτοιος χώρος που θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε τόσο για την εκπαίδευση, εκεί που δεν έχουμε κάνει, αλλά και για το διαδίκτυο. Και να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε μια κατάσταση στην οποία όλα θα είναι διαθέσιμα επιγραμμικά στο διαδίκτυο μέσω ψηφιοποίηση. Καλό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους εμπλεκομένους να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε τα πολιτιστικά ιδρύματα, τα μουσεία να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς να ποδοπατήσουμε τα δικαιώματα των κατόχων αλλά να μην αποκλείσουμε όλο αυτό το περιεχόμενο από το κοινό. Αυτή τη στιγμή, όπως σας προείπα, η ψηφιοποίηση βρίσκεται ακόμα σε εμβριακό στάδιο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Να σας δείξω και τα ακόλουθα δεδομένα. Όταν ζητούμε από τους κατόχους των δικαιωμάτων αν θα μας ε, έδιναν άδεια να χρησιμοποιήσουμε ένα έργο για το, για το άλλο, κάτι το οποίο είναι και δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αν λοιπόν τους ρωτούμε αν θα μας χορηγούσαν άδεια, η απάντηση δυστυχώ είναι κυρίως αρνητική. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να μιλήσουμε και με τον καλλιτέχνη και με άλλους. Στην περίπτωση που το έργο φιλοξενείται ας πούμε σε ένα μουσείο όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Κανονικά αυτό θα πρέπει να είναι πολύ πιο εύκολο. ήρθε υποτίθεται να πω και δύο λόγια την Ευρωπαϊκή, η οποία θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Όπως ακριβώς φαίνεται ένα έργο στο Ρίξ Μουζέου, στον ιστότοπο του Βασιλικού Μουσείου της Ολλανδίας. Έτσι θα έπρεπε να είναι διαθέσιμε οι συλλογέ στο ευρύ κοινό. Ευχαριστώ πολύ στο... για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η τελευταία πληροφορία που μας δείξατε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί κατά τη διάρκεια κροάσεων είχαμε την ίδια, με την ίδια εντύπωση. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν έργο στο διαδίκτυο, ακόμη και αν δεν είναι να βγάλουν τίποτα. Είναι μια συζήτηση που επανέρχεται διαρκώς, το να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο πάντω θα είναι δύσκολο. Κυρία Αν Κατρίν Λορά, ερευνητρία του Max Planck στο Ινστιτούτο. Ε, γερμανικά, αγγλικά, τα αγγλικά. Πολύ ωραία. Καλημέρα σα. Σας μέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να προσφωνήσω εξέχους, εξέχουσες προσωπικότητες σε, σε αυτή την συνάντηση. Από πλευρά ε, του Ινστιτούτου Ιδρύματος Max Planck ε, για τα πνευματικά δικαιώματα είμαι εδώ όμως ε, για να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις. Ενημερωτικά έχω συντάξει ένα πιο εξειδικευμένο έγγραφο το οποίο θα είναι η βάση ακριβώς αυτής της παρέμβασής μου και που είναι διαθέσιμη, στη, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ε, Επιτροπής σας. Πολλές ευκαιρίες, πολλές υπάρχουν για πρόσβαση στο διαδίκτυο για περιεχόμενα πολιτισμικού χαρακτήρα. Περισσότερες δυνατότητες από ό,τι φαντάζεται κανείς. Πρέπει να τα χειριστούμε και να τα προσανατολίσουμε σωστά. Όταν οι νομοθέτες και οι υπεύθυνοι για τις πολιτικές ε, ασχολούνται με αυτά, το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές ε, μια κατάσταση που ε, οδηγεί σε αδιέξοδο και αυτό όχι μόνο σε σχέση με την ε, ε, σκοπιμότητα ή όχι αλλά και επειδή είναι πολλές φορές ανεδαφικά τα μέτρα όταν μια νέα δυνατότητα για πρόσβαση ταυτοποιείται στην αγορά ως ευκαιρία για την αγορά οι νομοθέτες αρχίζουν να ασχολούνται στο να υπάρξουν συστήματα που θα οδηγούν στην προσαρμογή του, της νομοθεσίας στα νέα αυτά μέσα. Πολύ καλά. Αυτή είναι η ιστορία του, της προστασίας του copyright των πνευματικών δικαιωμάτων ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να δούμε τη σωστή εμβέλεια και εύρος. Φτάσαμε σε ένα κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη της, πληροφορίας, της κοινωνίας της πληροφορίας όπου θα πρέπει όχι να ρυθμίζονται από συμφέροντα της αγοράς στα θέματα πρόσβασης, αλλά θα πρέπει να διευκολύνονται από την ίδια την νομοθεσία για το copyright. Δεν μπορεί ο νόμος να είναι απλώς ένας ε, ακόλουθος ή εκτελεστής. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτι παραπάνω από ένα νομικό κείμενο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα με αρχές που θα είναι αρκετά στεναρές, ώστε να δίνουν ευκαιρίες ε, για πρόσβαση κάθε φορά που θα είναι προς όφελος των ε, ε, ατόμων και προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας συνολικότερα. Τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να αναγνωρίζουν την αξία της πρόσβασης σε σχέση με ένα πρότυπο αγοράς. Η ευρωπαϊκή πολιτισμική πολυμορφία είναι ένας τέλειος καταλήτης για την εσωτερική αγορά, για τα ωφέλη μια τέτοια χημική αντίδρασης. Και αυτή η χημική αντίδραση θα πρέπει να οδηγεί σε, από την ρύθμιση ενός ε, προτύπου ιδιοκτησία σε ένα πρότυπο πρόσβασης. Και σε σχέση και με τις ε, οργανώσεις καταναλωτών για τις οποίες είχα ε, εργαστεί. Με ρώτησαν συνάδελφοι Πώς μπορείτε να εργαστείτε για ανθρώπους που θέλουν όλα να τα έχουν δωρεάν στην πρόσβασή τους ε, όταν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ερώτηση είναι πώς ε, μπορεί κανείς ε, να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο για την βιομηχανία, για τα συμφέροντα των βιομηχανικών κύκλων. Δεν είναι δυνατόν να είναι αντιφατικές αυτές οι σχέσεις και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια σύνθεση. Ας πάρουμε το παράδειγμα σε σχέση με το cloud computing η νομοθεσία για το copyright όπως έχει σήμερα δεν διατυπώνει τις σωστές ερωτήσεις. Το θέμα δεν είναι να ξέρουμε αν και πώς τα δικαιώματα αναπαραγωγής ε, θα υποστούν ε, κάποιες επιπτώσεις από τις υπηρεσίες cloud computing. Φυσικά θα υπάρξουν τέτοιες επιπτώσεις. Το ερώτημα όμως είναι να αποφασίσει κανείς να επιτρέψει την πρόσβαση και τις ευκαιρίες ε, για τέτοιες υπηρεσίες που θα πρέπει να μπορέσουν να αναπτυχθούν ταχύτατα, χωρίς να χάνουμε χρόνο και σε σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές αξίες να μην χάνουμε χρόνο όσον αφορά και τις λεπτομέρειες, διότι γνωρίζοντας πώς τα δικαιώματα αναπαραγωγής ε, μπορούν να υποστούν επιπτώσεις ε, για την ευρωπαϊκή αγορά που θα είναι σημαντική και για να μπορέσουν οι χρήστες να μπορέσουν να υποφεληθούν από νέες καινοτόμες υπηρεσίες, που δεν σημαίνει ότι τα δικαιώματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να απολεστούν ή να μην προστατεύονται, αλλά όχι όμως σε ένα πολύ περιοριστικό πλαίσιο με πάρα πολλούς περιορισμούς. Ένα ανοιχτό πρότυπο πρόσβασης είναι συμβατό πρέπει να δούμε, που θα εστιάζεται στην πολιτισμική πολυμορφία και το πολυσχηδή χαρακτήρα της, προς όφελος των ε, ίδιων των πολιτών. Ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί δεν υπάρχει μια ανταλλαγή ε, όσον αφορά προϊόντα ε, μουσικής ε, στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα που όσον αφορά τέτοια φωνητικά προϊόντα, μουσικά προϊόντα, θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες τους. Αυτό για πολλούς λόγους. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ, ο Ευρωπαϊκός νόμος δεν προβλέπει άδειες για τέτοιου είδους ε, ε, διάχυση αυτών των προϊόντων στο διαδίκτυο. Στην Ευρώπη αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι δυνατό, θα μπορούσε. Αλλά πολλή δουλειά πρέπει να γίνει για να επιτραπεί κάτι τέτοιο και να μπορέσει να λειτουργήσει. Πρώτον, το καθεστώς όπως ισχύει σήμερα για το copyright θα πρέπει να μετεξελιχθεί και να μετεξελιχθεί σε ένα πλαίσιο πιο ευέλικτο, πιο ελαστικό. Αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία εξακολουθούν να είναι το πρότυπο θα πρέπει να είναι λιγότερο αποκλειστικά. Χρειάζονται περισσότερες εξαιρέσεις σε αυτό το στεγανό πλαίσιο. Και το ταμπού των υποχρεωτικών εξαιρέσεων πρέπει και αυτό να έρθει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα των εξαιρέσεων αποκλειστικά. Κάποιοι χρήστες θα πρέπει να μπορούν υπό πιο ελαστικούς όρους και προϋποθέσεις να έχουν ε, πρόσβαση σε θέματα ε, αναπαραγωγής και απομίμησης ε, τέτοιων προϊόντων. Όσον αφορά και την ερμηνεία, την εκτέλεση τέτοιων προϊόντων και να δούμε αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα με ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, copyright το που δεν πρέπει να κατακαιρματιστεί μεταξύ 27 κρατών μελών. Διπλασιάζεται αυτός ο κατακαιρματισμός από την έλλειψη ελαστικότητας μεταξύ των καθεστώτων που ισχύουν στα κράτη-μέλη, στα 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να μειωθεί αυτός ο κατακαιρματισμός και να υιοθετηθεί μια σφαιρική, συνολική πολιτική, ολιστική πολιτική για την ενοποίηση και όχι αποκλειστικά εναρμονισμό σε σχέση με κάποιες άκαμπτες διατάξεις. Αυτή η ελαστική πρόσβαση και αυτό το ελαστικό πλέον πλαίσιο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ελεύθερη πρόσβαση σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο συμφερόντων ε, κατέρωθεν. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα για το streamline στην Ευρώπη είναι το ότι το σημερινό σύστημα δεν επιτρέπει μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό οδηγεί στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα μελλοντικό τέτοιο πλαίσιο που θα πρέπει να ισχύει στην Ευρώπη σε σχέση με τους κανονισμούς αυτούς. Και αυτό έχει τη μεγάλη σπουδαιότητά του και σε σχέση με όρους πρόσβασης όσον αφορά υπηρεσίες που θα παρέχονται. Το σχέδιο οδηγίας για την συλλογική διαχείριση θα διαδραματίζει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις υποχρεώσεις ε, των εμπλεκόμενων, των παρόχων να δίνουν πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά τους στους για να μην δημιουργηθούν προβλήματα τροχοπέδησης όσον αφορά για παράδειγμα προϊόντα ε, που θα μπορούσαν να ε, δημιουργήσουν προβλήματα μέσω ενός άκαμπτου καθεστώτος θέματα τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα. Πρέπει να σκεφτούμε για μια καλύτερη κατάσταση, να μπορούμε με ευκολότερο τρόπο να ταυτοποιούμε τα δικαιώματα των χρηστών και να απλουστεύσουμε τα πρότυπα για την αδειοδότηση, για την χρήση τέτοιων δικαιωμάτων. Και υπό αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να έχουμε την καταχώρηση και τις ε, διευρυμένες, ε, ας το πω ε, για την αδειοδότηση. Αυτά θα δώσουν δυνατότητα να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τα πολιτισμικά θέματα και ένα ευρύτερο πλαίσιο για αυτές τις προσφορές. Κάτι διαφορετικό από το να προάγονται νομικές προσφορές ή δυνατότητες μόνο. Εδώ θέλω να εστιάσω την προσοχή σε ένα θέμα το οποίο δεν πολύ συζητήθηκε προηγούμενα και που πιστεύω εγώ ότι εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, να μην στρεβλωθεί η συζήτηση. Πρόσφατα βλέπουμε πολλούς πολιτικούς και ρυθμιστές να προάγουν τις legal offers, νομικού χαρακτήρα προσφορές ε, για την αντιστάθμιση ε, κάποιων άλλων μέτρων, δηλαδή μέτρων διαβαθμισμένων μέτρων για παράδειγμα, graduated ε, measures. Ως πραγματογνώμων για τα νομικά δεν γνωρίζω τι θα πρέπει να είναι ή τι είναι μια τέτοια νομική προσφορά, legal offer. Ε, εστιαζόμενοι στο παράνομο περιεχόμενο είναι πάντα η λάθος προσέγγιση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό ε, συνεπάγεται τον κίνδυνο να ε, έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές online, στο διαδίκτυο και να δημιουργείται αβεβαιότητα νομική και ανασφάλεια νομική. Τώρα θα πρέπει να εστιαζόμαστε στις ευκαιρίες περισσότερο, ευκαιρίες για την πρόσβαση και ακόμα για εκείνες που ακόμα δεν είναι εφικτές διότι θα πρέπει να δούμε τις αλλαγές και τις μεταβολές που είναι απροσδόκητες και δεν μπορούν όλες να προβλεφθούν και πρέπει να προσαρμοστούμε στο πλαίσιο αυτών των νέων ευκαιριών. Καθώς επίσης και για το εύρος των μη εμπορικών χρήσεων που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν ή συλλογικά να χαρακτηριστούν ως παράνομες. Μια τέτοια κατάσταση είναι αφόρητη για ε, όσους ε, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και θα μπορούσαν αυτοί δυνάμει, να, είναι, ε, να κάνουν καταχρηστική χρήση δικαιωμάτων ή να ε, ακολουθούν παράνομες ε, δραστηριότητες μέσα σε ένα τέτοιο ε, περιορισμένο πλαίσιο με περιορισμούς. Θα ήθελα να εστιαστώ σε μια άλλη πτυχή. Πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα και η αναθεώρηση το της οδηγίας για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα αυτού του πλαισίου. Κάτι όμως γίνεται για την πρόσβαση αυτού που θα πρέπει να γίνει και να, έχει πρόσβαση, να υπάρχει πρόσβαση για όλους. Ο δημόσιος τομέας που πρέπει να προστατεύεται από την ομοθεσία. Κάτι που αξίζει ως αγαθό να τύχει προστασίας. Είναι κάτι παραπάνω λοιπόν από ε, όλα τα άλλα θέματα, αυτός ο δημόσιος ε, χαρακτήρας, public domain. Το public domain, το, η δημόσια αυτή, το δημόσιο συμφέρον πρέπει να τύχει της προσπασίας. Πράγμα το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και οι Ευρωπαίοι νομοθέτες θα πρέπει να καταδείξουν την πορεία, τον προσανατολισμό που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Ja, ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο προβληματικό, πρέπει να πω. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση εδώ ενώπιόν μας που δεν είμαστε κράτος εμείς, είμαστε μια ένωση κρατών, 27 κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό το οποίο υφίσταται και είναι δεδομένο και το οποίο δεν ισχύει για τόσα πολλά χρόνια στα διαφορετικά κράτη να το εναρμονίσουμε με τέτοιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικίνδυνος όρος, όρος εναρμονισμός. Διαφορετικά όμως αν δεν προβούμε σε εναρμονισμό δεν θα είμαστε εταίροι των άλλων υπήρων της, ε, των ΙΠΑ, της Ασίας και άλλων και θα έχουμε διαρκώς προβλήματα. Ευχαριστώ για αυτές τις προτάσεις και ιδέες και για αυτό το θετικό συμπέρασμα στο οποίο οδηγηθήκατε. Προστασία του δημόσιου χώρου, public domain. Και θα λάβει τον λόγο τώρα στη συνέχεια από ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Humboldt. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Αγγλικά κι εγώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να απευθύνω τον λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην πρώτη μου διαφάνεια, όπως βλέπετε, έχω προσθέσει το ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό λογότυπο. Θα μιλήσω ως εμπλεκόμενο στην Ευρωπαϊκή από καταβολών του θεσμού. Μίλησα μάλιστα με το γραφείο μας στη Χάγη για να επικυρώσω το περιεχόμενο της παρουσίασής μου, αν και εκπροσωπώ τον εαυτό μου και μόνο στην ομιλία αυτή. Πέρα από, πέρα τα πραγματικά δικαιώματα υπάρχουν και, ξέρετε, τεχνικά ζητήματα που εμπλέκονται εδώ και τα οποία περιπλέκουν να περαιτέρω το θέμα. Δύο πράγματα λοιπόν θέλω να πω καταρχήν. Θα μιλήσω για την ψηφιοποίηση και την πρόσβαση και το που βρισκόμαστε ως προς τα δύο αυτά θέματα και θα μιλήσω επίσης για τα λεγόμενα linked open data και, τον, και το Google, τον περίφημο ελέφαντα στην αίθουσα αυτή που δεν βλέπει κανείς. Πρώτον, ψηφιοποίηση και πρόσβαση. Η πνευματική μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι ψηφιακή και σε ποιο βαθμό. Υπάρχει φυσικά η Ευρωπαϊκή Έχουμε και μερικά πολύ ενδιαφέροντα νούμερα εδώ, τα οποία δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 22 εκατομμύρια αντικείμενα στην Ευρωπαϊκή, 22 εκατομμύρια, πολλά από αυτά από την Γερμανία. Η κατάσταση ήταν διαφορετική μάλιστα πριν από λίγα χρόνια ως προς τα νούμερα. Πάντως το μεγαλύτερο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν υπάρχει εδώ. Φιλοξενείται όμως με τέτοιο τρόπο για τις ταινίες, με τέτοιο τρόπο όπως βλέπετε εδώ, όσον αφορά τις εφημερίδες ή κάπως έτσι όσον αφορά τα βιβλία. Ή σε ένα χάος σαν αυτό εδώ, το οποίο υποτίθεται ότι αποτελεί αρχείο. Η Ευρωπαϊκή, σε σύγκριση με όλα αυτά, ξαφνικά σας φαίνεται ένα πολύ μικρό κομμάτι. Ένα βασικό ζήτημα λοιπόν είναι πώς από την μικρή αυτή Ευρωπαϊκή θα οδηγηθούμε σε κάτι το οποίο θα είναι τουλάχιστον 10 φορές πιο μεγάλο. Οι αριθμοί για να καταλάβετε την κατάσταση υπάρχουν σε μια έκθεση που σας συνιστώ να διαβάσετε. Είναι προϊόν του έργου Enumerate. Και εδώ πάλι δεν μπορείτε να διαβάσετε τα στοιχεία αυτά, αλλά ε, μας λέει το διάγραμμα αυτό ότι όσον αφορά τα μουσεία δεν είμαστε και σε άσχημη κατάσταση. 42% του περιεχομένου έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Οι εθνικές βιβλιοθήκες όμως είναι στη χειρότερη θέση με ένα ποσοστό ψηφιοποίησης μόνο 4% του συνολικού περιεχομένου. Οι εθνικές βιβλιοθήκες έχουν πολύ δρόμο προφανώ μπροστά του. Επίση, το ήδη ψηφιοποιημένο περιεχόμενο δεν περιέχεται στην Ευρωπαϊκή. Μόνο 15% αυτού παρέχεται μέσω Ευρωπαϊκή. Παρά το γεγονό ότι η δυνατότητα υπάρχει. Και έχουμε και το θέμα βεβαίω τη ποιότητα τη ψηφιοποίηση. Ένα μεγάλο μέρο του υλικού έχει ψηφιοποιηθεί με τρόπο τέτοιο που σημαίνει ότι θα πρέπει να το επαναψηφιοποιήσουμε σε λίγα χρόνια. Πρόκειται δηλαδή για εικόνες που δεν είναι αξιοποιήσιμες τουλάχιστον για τους ειδικού και τους επιστήμονες. Έχουμε λοιπόν το θέμα της ψηφιοποίησης, το θέμα της ποιότητας της ψηφιοποίησης και το θέμα των μεταδεδομένων. Προαπαιτούμενο για την οποιαδήποτε αξιοποίηση. Θα σας συνιστούσα να κάνετε ό,τι μπορείτε για να προωθήσετε επενδύσεις στον τομέα αυτών, στην ψηφιοποίηση δηλαδή, και να ενθαρρύνετε, να παροτρύνετε τους εμπλεκόμενους να χωρίσουν περιεχόμενο, ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή. Επίσης, όσον αφορά την ε, ποιότητα της ψηφιοποίησης, χρειαζόμαστε τα λεγόμενα ανοιχτά πρότυπα. Γιατί πολλές φορές το περιεχόμενο ψηφιοποιείται με τρόπο τέτοιο, ώστε μπορεί να αξιοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί με ιδιόκριτα εργαλεία, τα οποία δεν είναι προσπελάσιμα στους περισσότερους χρήστες. Και εδώ ερχόμαστε στο σημαντικότερο ζήτημα. Linked Open Data. Ίσως να γνωρίζετε τα LOD από τις συζητήσεις που έγιναν στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την ενημέρωση στην δημόσια σφαίρα. Ο τρόπος διάθεσης του υλικού αυτού είναι το LOD. Ο Tim Berners-Lee τα είχε πει αυτά πριν από λίγα χρόνια, ο δημιουργός του διαδικτύου, Είπε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε δημόσια διαθέσιμα πρότυπα εργαλεία, εργαλεία αναγνώρισης, εργαλεία καθοδήγησης, εργαλεία συνδέσμων, ερωτήσεων και δηλώσεων στο διαδίκτυο στην αναζήτηση των δεδομένων. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτό, ειδού μια διεύθυνση στο διαδίκτυο, και υπάρχει ένα άλλο βιβλίο, ειδικά για την πολιτιστική κληρονομιά που δημοσίευσε ένας άλλος οργανισμός και υπάρχει και μια περίληψη για τους υπεύθυνου του τομέα. Στην Ευρωπαϊκή εμείς ακολουθήσαμε τον δρόμο του LOD. Εδώ έχω μερικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς έχουμε διαρθρώσει την Ευρωπαϊκή. Αυτά είναι LOD γραφήματα. Το μοντέλο που εφήβραμε για την Ευρωπαϊκή είναι ένα διαστρωματωμένο μοντέλο με αναπαραστάσεις αντικειμένων οργανωμένων σε αυτό το σύννεφο. Το σύννεφο αυτό περιέχει 500 δισεκατομμύρια περίπου δηλώσεις. Εδώ υπάρχουν όλο και περισσότερες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες και αυτό το έχει κάνει η Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή είναι κάπου εκεί πάνω δεξιά, αυτό είναι το, το σχετικό της μέγεθος. Και έχουμε και αυτόν τον μεγάλο πρωταγωνιστή να πως αποτύπωσε την ε, Google, το αλυσοδεμένο ποντίκι, το κανένα Σενέ στη Γαλλία. Και αυτή είναι η εκδοχή του Ζανουέλ Ζανενέ, ο οποίος ε, μας λέει το Google προκαλεί την Ευρώπη. Έπεισε έτσι έξι Ευρωπαίους ηγέτες να παροτρινούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει δήλωση για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με την παροκρουσίες το οποίο ήταν χρήσιμο γιατί άνοιξε τον δρόμο. Σήμερα έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι διαθέσιμο πάνω στο πρότυπο LOD, Linked Open Data. Πρόσφατα ξεκίνησε και αυτό το οποίο το Google ονομάζει The Knowledge Graph, το γράφημα της γνώσης. Πρόκειται και πάλι για διασυνδεμένε πληροφορίες, LD, αλλά δεν είναι ανοιχτό, δεν είναι προσπελάσιμο. Διότι το Google πήραξε λίγο το πρότυπο, έτσι ώστε η πρόσβαση να είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη. Το ερώτημα είναι, πρόκειται για μια διαφορετική εφαρμογή linked data. Όχι. Επίσης, μια άλλη πρωτοβουλία του Google, του Bing και του Yahoo και του Yandex η οποία λέγεται Είναι η προσπάθεια δημιουργίας ελεγχομένου λεξιλογίου για την περιγραφή και την αναζήτηση πολιτιστικών αντικειμένων στο διαδίκτυο. Είμαστε πολύ κοντά στο Link Data, στο πρότυπο του Link Data, όμως εδώ και πάλι υπάρχει προσπάθεια να πειραχθεί το πρότυπο και να περιοριστεί η πρόσβαση. Τα θέματα λοιπόν τα οποία οι πολιτικοί πρέπει να έχουν στο μυαλό τους είναι τα εξή. Τα linked open data και το γράφημα της γνώσης είναι φίλοι ή ανταγωνιστές. Τα LOD και η πρωτοβουλία σχήμα.org είναι συμπληρωματικές ή ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες. Και για μας η Ευρωπαίνα, την Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή και το Google πρέπει να συνεργαστούν υπό όρους, υπό ποιους όρους και σε ποιο βαθμό και με ποιες προϋποθέσεις. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να αποφασιστούν διότι έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν παράξενο παίκτη. Πρέπει να φροντίσουμε όμως να μην περιπέσουμε σε μια κατάσταση παράνοιας και η παράνοια είναι πολύ κακή όταν πρέπει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις. Θα συνιστούσα, αν μου επιτρέπετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσουν ε, μια πολιτική θέση όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να πείτε εσείς πώς βλέπετε το Google στο γενικότερο αυτό πλαίσιο. Θα ήταν χρήσιμο ίσως να πάρετε την γνώμη των ειδικών, θα συνιστούσα, θα σας προέτρεπα να δημιουργήσετε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα μπορούσε να συμπληκθεί σε συνεργασία με την Κομισιόν για να ρίξει μια πιο ενδελεχή ματιά σε μεγαλύτερο βάθος σε αυτήν την κατάσταση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά Γραμμάν. Λοιπόν, τέσσερις πραγματογνώμονες ακούσαμε στα όσα μας είπαν. Και μας δίνουν αρκετά, αρκετή τροφή με προτάσεις που σίγουρα κάτι μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτές, αλλά μας αφήνουν και πολλά ερωτηματικά εξίσου επίσης που πρέπει να ενασχοληθούμε με την απάντηση αυτών των ερωτήσεων και ερωτηματικών και να τα αναζητήσουμε αυτά ως απαντήσεις με ένα μέσο που θα μας βοηθήσει ώστε αυτά τα προβλήματα να μπορέσουμε με σοβαρό κάπως τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε και με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Ελπίζω ότι στη συζήτηση κάποια από αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Κύριε Μπόρις, έχετε τον λόγο. από την Πολωνία. Μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους πραγματογνώμονες. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα το πώς παρουσίασαν τα προβλήματα από τα όσα ακούσαμε. Τώρα έχουμε την εξή περίπτωση ως θέμα. Ουσιαστικά είναι κάτι το παράλογο αφενός. Διότι βλέπουμε ότι αφενός έχουμε μεγάλες προσδοκίες των πολιτών μας στην Ευρώπη. Των καταναλωτών και καταναλωτριών, των νέων. Μεγάλες προσδοκίες. Για όλους αυτούς το διαδίκτυο είναι ένα θεμελιώδου σημασία ε, μέσο όταν αναζητεί κανείς πληροφορίες. Είναι ο άτυπος τομέας μόρφωσης. Αυτός μορφώνει τους πολίτες. Το διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα νομικό και υποδομών που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πιστεύω ότι στις τεχνικές και τεχνολογικές, ε, στους τεχνολογικούς προβληματισμούς βέβαια, πρέπει να επιταχύνουμε την ψηφιοποίηση, οπωσδήποτε. Και όλα τα θέματα που συνδέονται με την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλειών και μέτρων, παράδειγμα, για ε, ε, Ευρωπιάνα, η πολυμορφοποίηση, κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων, προθεσμίες προγραμμάτων, χρονικά πλαίσια. Όλα αυτά πρέπει να είναι υπέρ της ψηφιοποίησης, να λειτουργήσουν υπέρ της ψηφιοποίησης. Έχουμε τα προβλήματα τεχνολογικά και τεχνικά την ενιοποίηση και εναρμονισμό που απαιτείται. Πρέπει τα κράτη-μέλη να ανεβάσουν ταχύτητα, να επιταχύνουν και να αναβαθμίσουν για να μπορέσουν να σημειωθούν πρόοδοι. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε το νομικό πρόβλημα. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν από την κυρία που παρενέβη, που είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο θάρρος περισσότερο θάρρος όσον αφορά την προστασία προς των πνευματικών ε, δικαιωμάτων. Ο κατακαιρματισμός που, ισχύει, που υφίσταται στην Ευρώπη με 27 διαφορετικά συστήματα, με εθνικούς φραγμούς και εμπόδια και προσκόμματα σε σχέση με τα πρότυπα τα οποία πορεύουν ιστορικά όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Είναι ένα μεγάλο εμπόδιο όλα αυτά. Ο κόσμος μεταβάλλεται άρδιν και ταχύτατα και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε με σταυρωμένα χέρια ως ε, θεατές αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να δράσουμε, να απευθυνθεί έκκληση, να επιταχυνθούν οι δραστηριότητες και οι δράσεις μας. Έχουμε ένα φως στην άκρη της σύραγγας που διαφαίνεται όσον αφορά όχι μόνο τα προϊόντα, προστασίας πνευματικών ε, δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια μικρή περίπτωση. Αυτά όλα τα νομικά θέματα σε ένα σφαιρικό πλαίσιο, όπως ε, η προστασία του κοινού ωφέλους και του δημοσίου συμφέροντος, public domain, πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη για να δράσουμε. Αυτή η ιδέα είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, το public domain ο δημόσιος χώρος και το κοινό συμφέρον για να δημιουργηθεί ένα πρότυπο ώστε σε αυτό το πλαίσιο να μπορέσουμε ευρύτερα στο διαδίκτυο να έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης και την δυνατότητα παρέμβασης των πολιτών. Σε σχέση με το Google δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ακόμα και σε, αν έχει κανείς αμφιβολίες, ξέρει κανείς τι γίνεται με το Google και την ψηφιοποίηση. Γνωρίζουμε τις εξελίξεις και σε σχέση με την ε, νομική επιτροπή και εκείνη ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά της ψηφιοποίησης και του Google Πιστεύουμε ότι εδώ χρειαζόμαστε, θα έλεγα, πώς να το πω, μια νέα τεχνολογία, χρήση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα επωφεληθούμε αυτών. Λοιπόν, με άλλα λόγια, για το public domain να μπορέσουμε να συνδέσουμε και να συνδυάσουμε αυτή την προσπάθεια προς προστασία του κοινού ωφέλους. Να υπάρξει ένα πρότυπο μιας SDIT, ε, δηλαδή μιας ιδιωτικής ε, και σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τα πράγματα και να δράσουμε αποτελεσματικά γιατί οι προσδοκίες των πολιτών μας είναι πολύ σοβαρές και ιδιαίτερα φιλόδοξες και αναμένουν οι πολίτες πολλά από εμάς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Παπα-Νικολάου από την Ελλάδα παρακαλώ. Και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και τους ε, εμπειρογνώμονες. Το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά την εισαγωγή σας και παρατήρησα ότι έχετε πολλά να μας πείτε σχετικά με την εμπλοκή του Google στη διαδικασία. Αν και γνωρίζω ότι το θέμα είναι υποσυζήτηση εδώ και πολύ χρόνο. Τελευταίος, προσφάτως, διαβάζω ότι το Google, το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται ταχύτερα στον τομέα αυτόν, το Google λοιπόν προτίθεται να προβεί σε ταχύτερη ψηφιοποίηση έργων εν γέννη και στην Ευρώπη σε πολλές περιπτώσεις ε, αγνοούν τα πνευματικά δικαιώματα. Ποια είναι η γνώμη σας περί αυτού, αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, εξίσου σημαντικό, στην προσφάτως ανακοινωθήσα στρατηγική υπάρχει πρόληψη να βρω το κείμενο και πείτε μου αν ισχύει όλο αυτό. Διαβάζω λοιπόν ότι αν και στην αρχή η διανομή θα είναι δωρεάν του περιεχομένου. Στο μέλλον θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τέλος πρόσβασης στα έργα. Ισχύει αυτό. Και έχετε κάποιο σχόλιο. ευχαριστώ. Η κυρία Βένα παρακαλώ, από τη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα βρισκόμαστε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ενδιαφέρον. Ε, οι εγκυκλοπαιδιστές ξεκινήσαν να κάνουν ένα ανάλογο έργο τότε. Δηλαδή να συλλέξει κανείς όλες τις πληροφορίες, τις γνώσεις και να τις προσφέρουν προς όλους. Βρισκόμαστε κάτι ανάλογο. Με ψηφιακό τρόπο πλέον. όπου θα έχουμε δηλαδή όλες τις πληροφορίες ψηφιακή πρόσβαση. Η κυρία Γκαλό στην Επιτροπή για τα νομικά είχε μια συνεδρίαση και υπήρξε πολύ ενδιαφέρον, ενδιαφέρον διάλογος, διότι υπάρχουν διαφορετικές προσέψεις. Ε, αυτά που είπε η κυρία Λορέν και σήμερα αυτό που διακυβεύεται είναι το εξή. Θα συνεχίσουμε με τα πνευματικά δικαιώματα όπως είχε μέχρι τώρα ή θα έχουμε το θέμα όπου έχουμε να κάνουμε μια κληρονομιά ή θα έχουμε μια πρόσβαση όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση σε, σε αυτά τα προϊόντα. Συζητάμε εδώ, προβληματιζόμαστε, διότι αυτά εδώ διακυβεύονται και το θέμα είναι έχουν να κάνουμε το δικαίωμα δηλαδή του πολίτη στην πρόσβαση στα έργα αυτά με ψηφιακό τρόπο, πώς θα γίνει αυτό και ποια θα είναι η νομοθεσία, ποιο θα είναι το κείμενο το νομικό που θα έχουμε για να υπάρξει αυτή η εφαρμογή. Και, και εδώ αυτό είναι το κεντρικό θέμα το οποίο δημιουργεί τις διαφορετικές προσήγησεις όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτό εδώ το, το χώρο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ενοποίηση θα λέγαμε των κειμένων. Δηλαδή να υπάρξει μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, αλλά πρέπει. Τώρα, Όσον αφορά την εξαίρεση για τα πνευματικά δικαιώματα, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται πολύ στη Γαλλία. Έχουμε τι εξαιρέσει όσον αφορά το χώρο του κινηματογράφου και σε άλλου τομεί. Να μα πούνε λίγα παραπάνω εδώ οι εμπειρογνώμονε, Ποιε είναι οι πιθανέ εξαιρεσει. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ενδεχομένω ανάλογα με το ποιο χώρο μιλάμε για τα... τον κινηματογράφο Φερρυπίν. Ε, υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά το καλλιτεχνικό προϊόν, δηλαδή αν έχουμε με τις φωτογραφίες ή κάτι άλλο φέρει Τα θέματα δεν, το θέμα αυτό με τις εξαιρέσεις δεν είναι και τόσο απλό. Η κυρία Λορέν τώρα, η οποία μίλησε και αναφέρθηκε όσον αφορά το θέμα της προσέγγισης για μια απλοποίηση των μεθόδων. Θα μπορούσε να μας εξηγήσει τι ακριβώς, πώς ακριβώς το εννοεί αυτό το θέμα με την απλοποίηση για να υπάρχει μια πιο εύκολη πρόσβαση. Και τώρα, αναφέρθηκε η, Ευρωπαϊ... η Ευρωπαϊκή Εγώ θα ήθελα να πω ότι έχουν αναφερθεί πολλά πράγματα όσον αφορά την τεχνική, αλλά όταν βλέπει κανείς ε, τις ιστοσελίδες φερπιν του Λούβρου ε, αντιμετωπίζει κανεί μια κατάσταση στην οποία είναι σίγουρο ότι υπάρχει πολλά που μπορούν να γίνουν πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Παράντα, την Γαλλία, παρακαλώ. Merci, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε δημόσια. Ε, πώς να οργανώσουμε νομικά ένα σύγχρονο σύστημα και όσον αφορά εμένα υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία είναι επιθυμητά, υπάρχουν όμως και υποχρώσεις. Ε, είναι κρίμα, είναι θλιβερό που έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ όσον αφορά αυτό το θέμα. Διότι υπήρξαν και θα λέγαμε θεολογικές αντιπαραθέσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, αυτά περάσαν. Τώρα έχουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Δύο κατευθυντικές γραμμές θα ήθελα να αναφέρω και που οποίες περιορίζουν την δημόσια δράση. Η, η πρώτη. Δεν μπορεί να έχουμε μία πολιτιστική, θα λέγαμε πολιτική, ε, η οικονομία μπορεί να εξασφαλίσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα πνευματικά δικαιώματα. Και από τη στιγμή πάλι που δεν θα έχουμε πρόσβαση, δεν θα υπάρχει δημιουργία ε, πνευματικών προϊόντων. Επιμένω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το πνευματικό δικαίωμα πρέπει να διασφαλιστεί. Αυτό θα πρέπει να είναι βάση μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο από κάθε θεσμικό όργανο εξάλλου το έχει υπογραμμίσει. Αυτό το έχει υπερασπιστεί. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα ότι μπορεί να κάνουμε κάποιες ε, αλλαγές ε, στο πώς ακριβώς θα γίνει η συλλογή των ε, στοιχείων, πώς θα, γίνει, θα ρυθμίσει το θέμα των αμοιβών. Μπορεί κανείς να το οργανώσει αυτά πολύ καλύτερα, αλλά να μην ξεπεράσουμε την κεντρική ιδέα. Ότι ο δημιουργός πρέπει να αμείβεται. Τελεία Παύλα. Επίσης, μια, η δεύτερη τώρα κατευθυντήρια μου γραμμή που υπάρχει, έχει να κάνει με συνεργασία των δημιουργών και του νομοθέτη θα πρέπει να έχουμε έναν άξονα όσον αφορά την οικονομική πτυχή, η δεμή θα καθυστερήσουμε και θα μείνουμε πίσω πάνω σε αυτό το θέμα. Θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή άλλα κράτη, άλλα έθνη, τα οποία είναι πολύ πιο δυναμικά και πιο φιλόδοξα, όπως η Κίνα πάνω σε αυτό το τομέα. Τώρα, να αναφέρω δύο ιδέες πάνω σε αυτό το θέμα, που μπορούμε να δουλέψουμε σοβαρά πάνω σε αυτές. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι οι δυσκολίες των δημοσίων οικονομικών για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι δυσκολίες πρέπει να αποτελούν επιχείρημα, ένα βάσιμο επιχείρημα, να μην δώσουμε μια βοήθεια όσον αφορά το, την προσπάθεια της χρηματοδότησης για την ψηφοποίηση. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ε, της δημόσιας προσέγγισης μέσω χρηματοδότησης, μέσω δανειοδότησης ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό και εδώ είναι κάτι το οποίο είναι επιτακτικό για να περάσουμε στην ψηφοποίηση. Υπάρχουν ε, τόσοι και τόσοι τομείς και αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε μια χρηματοδότηση, μια πολιτική χρηματοδότησης ε, για να μπορέσουμε να περάσουμε στην ψηφοποίηση. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα τώρα να αναφέρω όσον αφορά τα οικονομικά είναι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τα μεγαλύτερα ψηφιακά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν ένα μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα. Ε, ε, υπάρχουν τα κέρδη που έχουν κάνει και αυτό το βλέπουμε ότι δεν το, δεν το βρίσκουμε σε ε, κράτη στα οποία υπάρχει μια σωστή θα λέγαμε ε, ε, φορολογική κατάσταση. Αντιθέτως βλέπουμε σε κράτη, σε έθνη στα οποία υπάρχει μια ε, πιο χαλαρή αντιμετώπιση. Γίνονται συζητήσεις Φερρυπίν με τις ε, αρμόδιες αρχές στην Αμερική και την προσπάθεια να γίνονται επενδύσεις για να αναπτυχθεί περισσότερο αυτός ο τομέας. Εγώ τώρα, ότι δεν θα έπρεπε να αποφύγουμε μια τέτοια συζήτηση, είναι σημαντικό για τις δύο-τρεις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου να δούμε το θέμα που έχει να κάνει με τη φορολογική θα λέγαμε ε, κατάσταση. Και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αφορά την ψηφοποίηση, να συνεχίσουμε και να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. δεν θα μείνουμε πίσω, διότι το μεγαλύτερο μέρος της ε, πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν είναι ψηφοποιημένο. Λοιπόν, περιορισμός όσον αφορά να στηρίξουμε το, τα δικαιώματα τα πνευματικά του δημιουργού και μετά να δούμε πώς μπορούμε δραστικά να επιταχύνουμε τη διαδικασία για να ξεπεράσουμε την καθυστέρηση στην οποία βρισκόμαστε. Μετά το μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ Ζαμαρή Καβάντα. Και εγώ έχω κάποιε ερωτήσει. Πρώτον, μια ερώτηση. Φορέσατε τα ακουστικά σα Εντάξει, ωραία. Πρώτα, μια ερώτηση λοιπόν προς εκείνους που είπαν ότι υπάρχουν τόσα πολλά ψηφιοποιημένα προϊόντα. Ο καθηγητής Γκράτμαν νομίζω το είπε. Αλλά δεν διαβιβάζονται περαιτέρω στην Ευρωπαϊκή. Είναι και αυτό ένα θέμα που συνδέεται με κονδύλια, με χρήματα ή σε τι οφείλεται αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Κάνατε λόγο και είπατε ότι πρέπει να προβληματιστούμε μια ομάδα να δημιουργηθεί προβληματισμού πώς θα επιτευχθεί η συνεργασία με το Google και πού και πώς ενδεχόμενα μπορεί κάτι τέτοιο να χρησιμοποιηθεί, μια τέτοια συνεργασία να διευρυνθεί ερωτώ με, διαρωτώ με πράγματι σε αυτόν τον τομέα πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε, να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Έχει άλλη προσέγγιση το Google και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να προβληματιστούμε σίγουρα αν θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, μόνο που το ερώτημα είναι μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, μια τέτοια ανάληψη πρωτοβουλίας. Μετά όσον αφορά τα έργα αυτά Είχα μια μακρά συζήτηση το Σαββατοκύριακο στο Πότσταμ και όσον αφορά και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων πολλές ε, διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν αλλά κατέστη σαφές πόσο χρειαζόμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη μέχρι επιτέλους να καταλήξουμε σε μια κοινή οδηγία και κατεύθυνση. Το θέμα του Μητρώου, του καταλόγου έργων ε, αντιμετωπίστηκε. Ξέρω ότι ήδη στην Γερμανία προβλέφθηκε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν μπόρεσε όμως να εφαρμοστεί επειδή αναμέναμε την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Ξέρουμε ότι με 27 κράτη-μέλη ΕΕ πολύ δυσχερέστερα μπορεί να συνεργαστεί για να πετύχει κάτι τέτοιο. Απαιτούνται μακρότατες συζητήσεις. Σε αυτόν τον τομέα όμως πιστεύω ότι όλοι πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνες μας οι πολιτικοί εκπρόσωποι δεν είναι μόνο οι εθνικοί ε, πολιτικοί εκπρόσωποι που ε, δημιουργούν πολλές φορές προσκόμματα. Δεν πρέπει να χάσουμε τη δυνατότητα τώρα να δράσουμε. Θα πρέπει να επιταχύνουμε και να προχωρήσουμε. Το αναφέρατε και εσείς και ο συνάδελφος Μπόρις εξάλλου. Και στον κύριο Καβαντά θα ήθελα να πω το εξή. <clears throat> Σημείωσα ότι ποτέ δεν γίνεται λόγος για τους χορηγούς, sponsors. Σίγουρα έχουμε πολλές δυνατότητες από ιδιώτες να έχουμε κάποια χρήματα, κάποια κονδύλια για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Φυσικά μόνο εθνικά μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Δεν νομίζω ότι ευρωπαϊκά μπορεί να επιτευχθεί. Μπορεί κανείς να φανταστεί και έχει γίνει ήδη ακριβώς για αυτά τα θέματα όταν πρόκειται για ψηφιοποίηση, όταν πρόκειται για πολιτισμικά θέματα και πολιτιστικά του παρόντος και του παρελθόντος να βρούμε χορηγούς χορηγούς στους οποίους πρέπει να απευθυνθούμε για να ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν. Θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα για μας που θα εγγράφεται και θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κάποια κίνητρα ώστε άνθρωποι, πολίτες που θα έχουν πραγματικά κύρος και ε, περγαμίνες να προσπαθήσουν να εξεύρουν τέτοιου είδους χορηγούς που θα αφοσιωθούν στην ψηφιοποίηση, θα ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση. Διότι δεδομένη τη κατάσταση που έχουμε εμείς εδώ, δεν μπορούμε να απαιτούμε υπερβολικά πολλά πράγματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ξέρουμε ότι τα κονδύλια για τον προπολογισμό σπανίζουν τόσο πολύ, είναι τόσο ε, περιορισμένα, που δεν είναι δυνατόν με, αυτό, με αυτούς τους περιορισμούς να ασκηθεί κάποια επιρροή. Σε σχέση για παράδειγμα με μια υπερχρεωμένη χώρα που αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα. Λοιπόν, Ευτυχώς δεν χρειάζεται να υπάρχουν εξοικονομήσεις τέτοιες ε, από πλευράς π.χ. της Γερμανίας και ελπίζω ότι θα δώσει παράδειγμα μια τέτοια στάση διότι η πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά μας πρέπει να μπορέσει να διασφαλιστεί. Θα φτωχύνουμε αν δεν προστατέψουμε και δεν διασώσουμε αυτή την κληρονομιά. Η κυρία Σάκε παρακαλώ έχει τον λόγο τώρα. Η κυρία Σάκε. Um, Ευχαριστώ πολύ. Οι εισαγωγικέ παρατηρήσει ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσε. Ευχαριστώ του ομιλητέ. Έχω ερωτήματα πέραν αυτών που έθεσαν οι συνάδελφοι. Η συζήτηση στην εποχή τη ψηφιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία αφορά σε πολλές περιπτώσεις σε οικονομικά επιχειρήματα αλλά και το δημοσίο συμφέρον. Κάθε φορά που μιλούμε για συλλογική διαχείριση, την άκτα, τα ορφανά έργα, ξέρουμε ότι εμπλέκονται σημαντικά λόμπι. Ακούμε τη φωνή των εκδοτών, των κατόχων των δικαιωμάτων, της μουσικής βιομηχανίας, των Οργανισμό Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματική Ιδιοκτησία. Και αυτέ οι φωνέ είναι πολύ πιο δυνατέ από τι φωνέ των μουσείων, των βιβλιοθηκών και του κοινού. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κέλλερ συγκεκριμένα, γιατί το ανέφερε στην ομιλία του, ότι κάποια μουσεία δεν θέλουν να διαθέσουν τα έργα του επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Και μια ερώτηση προ όλου του μιλητέ. Πιστεύετε ότι οι πολιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορεί ε, έχουν αντίστοιχε επιφυλάξεις πως πρέπει να θεσπίσουμε ρήτρες περαιτέρω ευελιξίας πριν μεταρρυθμίσουμε ριζικά εκβάθρον το σύστημα. Να εισαγάγουμε την έννοια της θεμητής χρήσης όπως στις ΗΠΑ, το fair use δηλαδή. Μήπως αυτό θα βοηθούσε. Και ξέρετε αν υπάρχουν μελέτες, αν έχει γίνει έρευνα σχετικά με το ποια είναι η βέλτιστη μεταρρύθμιση η οποία θα επιφέρει και τα μεγαλύτερα ωφέλη στην κοινωνία μας εν τέλει. Πιστεύετε ότι η φωνή των δημοσίων φορέων ακούγεται επαρκώς και φοβούμαι επίση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη εν γέννη χάνει έδαφο σε σχέση με τις ΗΠΑ διότι εδώ οι περισσότεροι ασχολούνται με την προστασία των δικών τους δικαιωμάτων και μένουν προσκολλημένοι στο παρελθόν. Οι κυβερνήσει δεν είναι στην εξουσία για να προστατεύουν υπέρμετρα τα πνευματικά δικαιώματα. Το είπε και ο Σάνφος ε, Μπόρις. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις δικές μας εσωτερικές αντιφάσεις και αντιμαχίε. και δεν έχουμε τελειώσει ως πως αυτό που είπε και ο κ. Καβαντά. Υπάρχουν σοβαρές ε, διαμάχες ακόμη και εντός του Κοινοβουλίου μεταξύ αυτών που είναι υπέρ της μεταρρύθμισης και αυτών που είναι υπέρ της διευρυμένης πρόσβασης. Χρειάζεται να δώσουμε στους δημιουργούς περισσότερες ευκαιρίες, αλλά πρέπει να αναθεωρήσουμε και τον ρόλο των κυβερνήσεων και μετά να δούμε τι θα κάνει και η αγορά. Στην ψηφιακή εποχή πρέπει τα πνευματικά δικαιώματα και ο τρόπος υλοποίησής τους δεν μπορεί να απαγορεύει, να δυσκολεύει και το να περιέλθουν τα κέρδη, το ωφέλη στους δημιουργούς. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη δημιουργών και του κοινού. Πρέπει λοιπόν τα επιχειρηματικά μοντέλα να προστατεύσουν αυτές τις δύο πλευρές κατά κύριο λόγο. Αλλιώς βρισκόμαστε σε μια ε, κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα ήθελα τις απόψεις για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εντάξει, η κυρία Μπέναραμπ Ατού, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε κύριο Καναντά, το θέμα για τα θέματα για το εισόδημα των δημιουργών είναι σίγουρο ότι αν δεν διασφαλιστούν αυτοί δεν θα έχουμε δημιουργία. Το, το ερώτημα. Αν λέμε ότι θα πρέπει τα έσοδα να πάνε στους δημιουργούς. Ε, έχουμε μια κατάσταση στην οποία ακόμα και αν πεθάνει ο, με αυτά που ισχύουν ο δημιουργός για 50, 60, 70 χρόνια οι κληρονόμοι ε, ε, δέχονται ε, εισοδήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο δεν έχουν δημιουργήσει. Υπάρχει δηλαδή το θέμα του δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων όσον αφορά τη διάρκεια. Και τώρα θα δώσω τον λόγο πάλι στους επαΐοντες, στους πραγματογνώμονες. Ποιος θέλει να ξεκινήσει παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε από τα δεξιά και πάμε αριστερά προς τα αριστερά. Ο κύριος καθηγητής Γκράτμαν. Αρκετές ερωτήσεις ε, μου απευθύνθηκαν. Ξεκινώ με το Google. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην παρουσίαση το Google θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό εταίρος σε αυτά τα οποία γίνονται. Πολλά σε σχέση με την ψηφιοποίηση που έχουν ήδη επιτευχθεί στην Ευρώπη έγιναν με βοήθεια του Google. Το πρόβλημα όμως ήταν σε σχέση με αυτή την πτυχή τώρα εδώ με το Google ότι ένας αριθμός θεσμικών οργάνων που γνωρίζω, για παράδειγμα η Βαβαρική Βιβλιοθήκη στο Μόναχο, η Εθνική Βιβλιοθήκη στη Βιέννη της Αυστρίας, έχουν συμβάσεις με το Google που πρώτον δεν είναι διαφανής, δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν οι όροι αυτών των συμβάσεων. Αυτό είναι κάτι σκανδαλώδε, πιστεύω εγώ στοιχείο. Και το δεύτερο είναι, και αυτό απαντά το θέμα της μη διαθεσιμότητας ψηφιοποιούμενων στοιχείων, Αυτές οι συμβάσεις φαίνεται ότι αποκλείουν το δικαίωμα της ελευθερίας αναδιανομής ψηφιοποιημένων προϊόντων και συνδεδεμένων metadata. Δηλαδή προφανώς δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο αυτών των συμβάσεων. Οι συμβάσεις συνάπτονται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή υπό τη σημερινή μας πολιτική. Για παράδειγμα, ότι όλα τα metadata θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα για καθέναν, για οποιαδήποτε χρήση. Και φαίνεται ότι υπάρχει εδώ μια αντίφαση, ένα, υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα εδώ. Είναι ένα νομικό ε, θέμα αυτό φυσικά αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε και να φροντίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα, θα ε, προβαίνουμε σε συμβάσεις με, το Google στο μέλλον. Πώς θα συνάπτονται αυτές οι συμβάσεις. Δεύτερον, το κοινωνικό όφελος, ε, public domain, το δημόσιο όφελος. Υπάρχουν μελέτες ε, και μελέτες που έγιναν υπό τη δική μου εποπτεία στο Βερολίνο, που μπορώ να διαθέσω βέβαια, γιατί πραγματικά πιστεύω και το προέβλεπα αυτό το ερώτημα θα ετίθετο. Εκτός αν είμαστε σε θέση να πούμε σε εσά και άλλους νομοθέτες και πολιτικούς στο άμεσο μέλλον τι είδους πρόσθετη αξία δημιουργείται από την Ευρωπαίανα και ποιου είδους αξία γίνεται με την μορφοποίηση αυτών των προϊόντων σε ψηφιοποίηση, θα υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν θέματα λοιπόν που είναι διαθέσιμα που όμως δεν έχουν προετοιμαστεί για, την, για ε, ελεύθερη χρήση από χρήστες, είναι ευρύτερες μελέτες, θα ε, έπρεπε να είναι, θα μπορέσουμε να σας τα διαθέσουμε για να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει σαφής τοποθέτηση για το πώς αυτά πρέπει να διαμορφωθούν και μπορεί λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη από εσάς, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να συνειδητοποιήσετε είναι είναι πολύ ισχυρό ε, παίκτη ω εμπλεκόμενο η Google. Εμείς στην Ευρώπη είμαστε και εμείς ισχυροί ε, πάροχοι και παίκτε. Το πρότυπο με την Ευρωπαϊκή, το τεχνικό αυτό πρότυπο, ε, βρίσκεται, έχει πρότυπο την ψηφιοποιημένη βιβλιοθήκη της Αμερικής. Έχουμε μία λοιπόν περίπτωση όπου είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη εμείς τεχνολογικά και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το μέσο όσο το έχουμε στη διάθεσή μας και να προχωρήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ως προς αυτό ότι το Google έχει ζωτικό συμφέρον να συναλλάσσεται και να διαβουλεύεται μαζί μας. Έχασαν την άβρα του μόνου ε, εμπλεκόμενου έχουν εμπλακεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊάνα για να αποκαταστήσουν το ε, προηγούμενο καθεστώς προπομπού που είχαν, αυτή την άβρα την οποία έχασαν εντωμεταξύ. Το τελευταίο θέμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την Ευρωπαϊάνα είναι ότι ναι, σε σχέση με αυτό που είπατε, θα το διαβιβάσω στη Χάγη την παρατήρησή σας. Μπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο ως προς αυτό που είπατε. Θα καθελκυστεί μια νέα τέτοια ε, πρόταση, διατύπωση το Νοέμβριο από πλευράς μας. Εργαζόμαστε με πρότυπα τα οποία είναι πολύ πιο διαδραστικά. Αυτό το οποίο λείπει στην Ευρωπαϊκή δεν είναι σε σχέση με κάποιες ε, μελέτες ή στοιχεία, είναι η διαδραστικότητα που απουσιάζει. Προσπαθούμε να δράσουμε και να λάβουμε μέτρα σχετικά. Γνωρίζουμε τις ελλείψεις ε, και τα μειονεκτήματά μας και πρέπει να τα αποκαταστήσουμε αυτά. Αυτά νομίζω είναι τα θέματα που αναφερθήκατε και έπρεπε να απαντήσω. Ευχαριστώ. Okay. Ε, ευχαριστώ. Εσείς κυρία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το γιατί η νομοθεσία δεν έχει ήδη προβλέψει κυρώσει, δεν έχει αντιμετωπίσει το φαινόμενο Google. Ε, κοιτάξτε, προς το παρόν η νομοθεσία αντιδρά κατά περίπτωση δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Απαιτείται χρόνος λοιπόν μέχρι να σχηματιστεί μια γενική εικόνα του φαινομένου. Γι' αυτό και πρέπει να δημορφώσουμε καταρχήν άποψη περί του θέματος και να ενσωματώσουμε το συμφέρον του κοινού στη συζήτηση και στην νομοθεσία. Αλλά αυτό δυστυχώς παίρνει χρόνο. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις όσον αφορά την νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα θέσπισης ε, τέλους πρόσβασης σε περιεχόμενο. Έχει συζητηθεί εκτενώς βεβαίως. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Υπάρχει πρόταση που αφορά την δημιουργική συμβολή, όπως λέγεται. Όλες οι λύσεις πάντως κατατείνουν προς την διαχείριση, κατά κάποιο τρόπο, τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Αλλά το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι υπάρχει αμοιβή εν τέλει. Σίγουρα πρέπει να γίνει περισσότερη συζήτηση και κάπου να καταλήξουμε, αλλά δεν ξέρω πού προς το παρόν θα καταλήξουμε. Όπως είπα και στην παρουσίασή μου, υπάρχουν λύσεις όπως η παράταση της συλλογική διαχείρισης, το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα ενδεχομένω λύση είναι λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς, ε, οι οποίες πολύ συχνά χαρακτηρίζονται ως οι σκανδιναβικές λύσεις. Στην Ορβηγία και στη Σουηδία έχουμε τέτοιου είδους συλλογικές άδειε, οι οποίες λειτουργούν ικανοποιητικά. Γιατί να μην επεκτείνουμε αυτές τις λύσεις, τις ήδη λύσεις, σε ένα ευρύτερο αντικείμενο. Είναι κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να δουλέψει. Τώρα, όσον αφορά τις εξαιρέσεις, θεωρώ ότι απαιτούνται ελάχιστα πρότυπα υποχρεωτικών όμως εξαιρέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτές οι υποχρεωτικές εξαιρέσεις θα υπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, όπως η εκπαίδευση, η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό στην αναθεώρηση τη οδηγία περί προστασία πραγματική διοκτησία μπορεί να ενσωματωθεί. Υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίω, αλλά χρειαζόμαστε κάποιου ελάχιστου κανόνε. Όχι μόνο για τι εξαιρέσει, αλλά και για τα μοντέλα επιτρεπόμενη θεμητή χρήση. Αν διαβάσετε την οδηγία περί ορφανών έργων, λέει για επιτρεπόμενη χρήση των ορφανών έργων. Στην πρώτη διατύπωση δεν προβλέπεται εξαίρεση στο κείμενο. Όμως τις ε, επακόλουθες εκδοχές του κειμένου το προβλέψαμε. Αν διαβάσετε πάντως προσεκτικά το κείμενο, όλα αυτά τελούν υπό πολλούς περιορισμούς και γι' αυτό ξαναλέω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία η έννοια της δημόσιας σφαίρας θα μας επιτρέψει να υπερβούμε τις δυσκολίες ε, και να αφήσουμε πίσω μας αυτό το μη ικανοποιητικό σύστημα εξαιρέσεων. Και προκειμένου ε, να πω κάτι για την παρέμβαση του βουλευτή από την Πολωνία. Και δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά πιστεύω ότι στην Πολωνία υπάρχει συγκεκριμένη προστασία της δημόσιας σφαίρας. Καθώς και παράλληλα αμοιβή γι' αυτό. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να εξετάσουμε την πολωνική λύση σε μεγαλύτερο βάθος. Τώρα η δημόσια σφαίρα, ο δημόσιος χώρος, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει ως έννοια, αλλά δεν είναι ένα ανοιχτό μουσείο με αξιοπερίεργα όπως λέμε. Δεν είναι το ντουλάπι με τα αξιοπερίεργα. Πάντως σίγουρα υπάρχει και πρέπει να προστατευτεί. Η δημόσια σφαίρα απορρέει, προκύπτει όχι μόνο από την εκπνοή των δικαιωμάτων, αλλά και από την εθελούσια προσφορά των δημιουργών να απεμπολίσουν τα δικαιώματά τους. Κάποιοι δεν θέλουν, δεν απαιτούν προστασία, δεν θέλουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Συνομολογούν δηλαδή την απεμπόληση των δικαιωμάτων τους και έτσι αυτά ανήκουν πλέον αυτομάτως στην δημόσια σφαίρα. Το επόμενο ερώτημα αφορά τον κατάλογο έργων, το μητρό έργων Το μητρό αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο από μια βάση δεδομένων που επιτρέπει πρόσβαση πληροφορίε σχετικά με τα έργα. Έτσι δεν θα έχουμε πλέον ορφανά έργα και θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά η αγορά. Είναι ένα καυτό βεβαίως θέμα και δεν αποτελεί σύμπτωση ότι η WIPO έχει ιδρύσει ομάδα εργασίας για να μην για τα μουσικά έργα. Ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια βάση δεδομένων έργων μουσικής. Αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα λύση. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, Κρετάλα, με την άλλη παρατήρηση που αφορούσε την απουσία του κοινού, της, δημόσιας, της κοινής νόμης από τη συζήτηση, από τον δημόσιο διάλογο. Έχω δει τη διαφορά. Όταν ε, δούλευα για τη μουσική βιομηχανία, για τον τομέα της μουσικής, ήταν πολύ πιο εύκολο να έχω πρόσβαση στους πολιτικούς. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Οπότε δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτό που είπατε. Και αν υπάρχει συνένεση, συμφωνία μεταξύ των ε, κατόχων δικαιωμάτων, ε, κοιτάξτε, εξαρτάται από τον τομέα. Είναι πολυτομιακή η προσέγγιση. Κάποιοι πιο δημιουργικοί τομεί δύσκολα έχουν κέρδη. Ας πούμε, οι εκδότες, ο τύπος, κάποιοι εκδότες του, τουλάχιστον. Η συζήτηση γίνεται όλο και πιο τομεακή. Οπότε είναι δύσκολο να εκφέρει κανείς γνώμη, άποψη για όλους τους τομείς μαζί. Χρειάζεται περαιτέρω εργασία. Ευχαριστούμε εσείς κύριε Κέλλερ παρακαλώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολλές ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές απαντήθηκαν ήδη από τους συναδέλφους μου μόλις πιο πριν. Επιτρέψτε μου να τις πάρω κάποιες από αυτές εξετάζοντας τις. Πρώτον, ο Ευρωβουλευτής από την Πολωνία σε σχέση με την οδηγία είπε «Βλέπουμε φως στο τέλος της, στην άκρη της σύραγγας». Τίνω να διαφωνήσω απόλυτα με αυτό, διότι η οδηγία για τα ορφανά μη προστατευόμενα αυτά προϊόντα δίνει κάποιες ευκαιρίες για, την, ε, για έργο από πλευράς μας. Αν δει κανείς τα θέματα, δηλαδή πρόσβαση σε orphan works, δηλαδή για την μη διαθεσιμότητά τους. Ε, είναι, ας το πω έτσι, ένα εγχείρημα για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, για την διατήρηση, διασφάλιση κάποιων αρχών που πρέπει να τηρηθούν. Καταλήξαμε σε μια λύση που θέτει το βάρος στα ιδρύματα που εργάζονται με κονδύλια, δημόσια κονδύλια, για να διασφαλιστεί αυτή η πτυχή. Δηλαδή, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με το ελάχιστο αυτό επίπεδο προστασίας για ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι θέμα κακής αρνητικής νομοθεσίας που δεν προέβλεψε αρχικά το ότι κάποτε θα ήταν διαθέσιμο το διαδίκτυο και δεν είχαμε το θάρρος να δραχθούμε τις ευκαιρίες και να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο και τις διατάξεις. Βρισκόμαστε λοιπόν υπό τον πριτανεύοντα ρόλο ε, όπως προαναφέρθηκε ότι Είμαστε όμοιροι σε καθεστώς ομοιρίας από ανεδαφικές διατάξεις, συμφέροντα τα οποία έχουν ήδη ε, αποκρισταλωθεί και που δημιουργούν ένα αρνητικό πλαίσιο εξισορρόπησης. Δεύτερη παρέμβαση που αναφέρθηκε σε σχέση με τον κύριο ε, Στέφαν Γκράτμαν. Παρότι συμφωνούμε με πολλές από τις επικρίσεις ε, που έγιναν, το Google πρέπει να το δούμε ως έναν εξαιρετικό εξαίσιο εταίρο για τις δυνατότητες που διανοίγονται. Σε σχέση με το συνέδριο για ε, ε, ένα Ιταλικό ε, μητρό το οποίο είχαμε με την ε, συλλογή ενός ε, συλλέκτη όχι μόνο στο YouTube που δημιουργεί πολλούς θεατές, μιλιάδες θεατές για αυτό το υλικό, πολύ περισσότερους από ό,τι αν παραμείνει κανείς σε μια στενή πλατφόρμα αρχικά, αλλά και σε σχέση και με την διαφήμιση και ε, το έργο που συνεπάγεται η δράση του Google με τα στελέχη του και τους υπαλλήλους. Αν δει κανείς το Google με όλα τα θετικά, πολλές υπηρεσίες παρέχονται από το Google που ουσιαστικά έχουν τεράστια αξία για ιδρύματα πολιτιστικής προστασίας κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι, μπορεί, μπορεί να είναι και είναι ένα σημαντικός εταίρος. Μπορεί κανείς να δει κανείς ε, και άλλες, ε, άλλα τέτοια εγχειρήματα, για παράδειγμα και καλή εκπροσώπηση και από πλευρά Ευρώπη που μπορεί να εξυπηρετούν το ίδιο, τα ίδια συμφέροντα, αλλά να μην τα βλέπουμε μαύρα άσπρα τα πράγματα με ακραίο τρόπο. Για τα ερωτήματα που απευθύνθηκαν σε μένα, πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να δομήσουμε τις εξαιρέσεις για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας τους. Δεν χρειάζονται εδώ περίπλοκα πλαίσια και περίπλοκες ρυθμίσεις. Δύο κύρια πράγματα. Πρώτον, για μια εμπορική χρήση, δημόσια διάθεση και ε, προσπελασιμότητα, χωρίς ε, να υπάρχουν προσκόμματα, να δείχνεται να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό το δημόσιο χωρίς περιορισμούς. Και για κάποιους ε, τομείς με συγκεκριμένα προβλήματα, εδώ θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή. Πώς θα κάνουμε, θα χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή σε σχέση με προϊόντα που βρίσκονται σε εμπορική εκμετάλλευση και την δυνατότητα χρηστών να μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς να υπονομεύονται αυτά τα ε, εμπορικά πρότυπα για την μεγάλη πλειοψηφία υλικού που δεν βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να επιληθούν τα προβλήματα. Σε σχέση με τα εμπορικά εκμεταλλευόμενα υπάρχουν τα θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας όπως προαναφέρατε. Δηλαδή ο δημιουργός πρέπει εκείνος ο οποίος πρέπει να δρέπει τα ωφέλη <clears throat> Αν όμως κανείς δεν είναι εκείνος ο οποίος ε, μπορεί να ε, αποκομίσει αυτά τα ωφέλη ως ε, κέρδος, ως έσοδα, τότε δεν πρέπει να περιπλέκονται τα πράγματα, ώστε να μπορέσει να αναζωογονηθεί ένα έργο ως προς το προσδόκιμο ζωής του και να αναζωογονηθεί σε σχέση με την προσπελασιμότητα, διαθεσιμότητα των χρηστών. Εδώ, σε σχέση με την ψηφιοποίηση και την πρόσβαση, εδώ είναι ένα, μπορεί να είναι περίπλοκο αυτό το θέμα ένα από τα θέματα που μάθαμε, από τα ζητήματα που είδαμε ήταν όταν ψηφιοποιεί κανείς χωρίς να έχει ρυθμίσει το θέμα της πρόσβασης εκ προημίου, καταλήγει κανείς σε μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογηθεί σε σχέση με την, το, αντίτιμο των κονδυλίων που χρειάζονται για την ψηφιοποίηση τόσων προϊό, τέτοιων προϊόντων όταν δεν μπορεί να υπάρξει όφελος με την ελεύθερη πρόσβαση για χρήστες. Θα πρέπει να βρεθεί μια αρχή που θα όταν θα ψηφιοποιούμε υλικό θα μπορεί να είναι διαθέσιμο στο δημόσιο, στους χρήστες δημόσια να μπορούν να, να δουν οι πολίτες την αξία των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την ψηφιοποίηση προϊόντων και τη βούλησή μας με τέτοιου είδους ε, προγράμματα να ε, είμαστε επωφελείς προς το ε, κοινό. Και δεύτερο ή εν τέλει το θέμα της ταχύτητας της νομικής ρύθμισης ειλικρινά αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα συζήτησης, αλλά δημιουργεί και πολλές ανησυχίες. Το ανέφερα σε σχέση με την ψηφιοποίηση ε, για την μελλοντική χρήση. Το YouTube δεν υπήρχε τότε. Κάνουμε λόγο λοιπόν για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν άλλαξε σημαντικά από το 2001 σε σχέση με τις αλλαγές που επήλθαν ε, ε, μεταγενέστερα και δεν βρήκαμε τρόπο να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια όσον αφορά το εύρος των προβλημάτων. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς μια νομική δομή που θα μπορούσε, ας το πω έτσι, να προβλέπει ένα νομικό χτένισμα ή σε τακτά πλαίσια προσαρμογών. Αν σκεφτεί κάποιος, για παράδειγμα, τον κατάλογο εξαιρέσεων που έχουμε, που πρέπει σε τακτά διαστήματα να επικαιροποιείται, να αναθεωρείται κάθε τέσσερα χρόνια π.χ. Ένα τέτοιο μηχανισμό να προβλέψουμε, ώστε να μπορεί κανείς να προσαρμόζεται στις αλλαγές ε, σε ε, μικρότερα διαστήματα, σε τακτά διαστήματα. Πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την ε, ταχύτητα των νομικών ρυθμίσεων και να μην αποβαίνει η κατάσταση αυτή εις βάρος του νομικού πλαισίου και των χρηστών. Και τέλος, για τα ερωτήματα από την κυρία Σάκε. Φοβούμαι ότι δεν υπάρχει πραγματική συνένεση από πλευράς του τομέα της προστασίας πολιτισμικής κληρονομιάς, τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Εδώ πρέπει να δούμε και τις δυνατότητες που έχουν οι εθνικές αρχές σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Αν ασκούν πίεση οι εθνικές αρχές για να υπάρχουν έσοδα σε σχέση με τη διάθεση τέτοιων προϊόντων στο διαδίκτυο, διαδικτυακά, τότε μπορεί κανείς να δει μια πολύ πιο συντηρητική προσέγγιση ή εγωιστική με την επιλογή του τι διατίθεται σε δημοσιογραφία δημόσια χρήση ε, για την αποκόμιση κέρδους. Αν δεν υπάρχει κάποια τέτοια περιοριστική προσέγγιση μπορεί κανείς να είναι πιο ελεύθερος ή φιλελεύθερος προοδευτικός και να έχει ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο που θα δημιουργήσει. Και πρέπει να δούμε στην ψηφιακή εποχή ότι υπό το δικό μου πρίσμα αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει το γεγονός ότι θα είναι διαθέσιμο το υλικό αυτό όσο το δυνατόν ταχύτερα προς το κοινό και αυτό ε, συνεπάγεται και τη συζήτηση σε σχέση με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αλλά πρέπει όλο και περισσότερο αυτές οι ενώσεις ε, να εμπλακούν και να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα για την τελευταία ε, ερώτηση για την χρήση για αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε περισσότερο ελαστικές διατάξεις όσον αφορά το copyright. Ίσως το πρόβλημα πρέπει να το δει κανείς ότι καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε θα πρέπει να ε, βρούμε τον ιδανικό τρόπο να επιληθούν τα προβλήματα και οι εξαιρέσεις ή τις τέσσερις αρχές ε, πρόσβασης, προσέγγισης. Αυτή η αρχή είναι αν δεν βλάπτει κάτι όσον αφορά τα υποκείμενα οικονομικά συμφέροντα, τότε θα μπορούσε να είναι θετική προσέγγιση. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να εμπνέει την νομοθεσία. Να δούμε πού γίνεται ζημιά, πού υπονομεύονται τα πράγματα. Και εδώ υπονομεύονται τα πράγματα όταν ε, επενδύουμε σε ψηφιοποίηση και δεν μπορεί να αποβεί προς το κοινό όφελος, ε, προς το όφελος των πολιτών. Πρόκειται για επένδυση από την οποία θα πρέπει να υποφεληθούν από αυτή την ψηφιοποίηση. Το να δίνουμε το ένα και να υπάρχει, ε, ας το πω έτσι, ένα αντίδωρο από την άλλη πλευρά. Ψηφιοποιούμε, αλλά προς το κοινό όφελος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός. Μάλιστα, θα είμαι πολύ σύντομος διότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα χρονικά όρια. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν νεότερες, νεότερες εξελίξεις. Νομίζω κοιτάζουμε τα θέματα παραδοσιακά και παραβλέπουμε ότι αυτά τα οποία γράφουν σήμερα την ιστορία είναι τα τεκτενόμενα, οι επαναστάσεις που συμβαίνουν και στον ιδιωτικό μας χώρο βλέπουμε ότι έχουμε κατακλυσμό, κατακλυσμό που, μας, που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το facebook ή τα κοινωνικά μέσα, social media. Ερωτώ, ποιος είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να πει ποιος είναι αρμόδιος τελικά και τελεσίδικα για όλα αυτά. Δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ όπως για του τηλεοπτικού σταθμού πριν από 30 χρόνια είχαμε μια τέτοια ε, ένωση, ένα τέτοιο σώμα για παράδειγμα. Σήμερα έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο. Τα νέα κοινωνικά μέσα. Πού θα βρεθεί η αρμοδιότητα για αυτά σήμερα. Ενώ εμείς ασχολούμαστε με όλα αυτά τα ανεπίλητα θέματα, copyright και όλα αυτά τα, ας το πω έτσι, ε, από το παρελθόν που έχουμε κληρονομήσει αν βλέπουμε ότι τότε δεν υπήρχαν σαφή νομικά πλαίσια το παλαιό δεδομένο ε, μια νυχτή θα έπρεπε να είχε απελευθερωθεί. Δεν, έγινε, δεν, αυτό. Το δεύτερο είναι ποιος θα ενδιαφερθεί για τους ιδιωτικούς, ε, τα ιδιωτικά κανάλια τηλεοπτικά. Πουθενά δεν υπάρχει, ας το πω έτσι, η ε, αναγκαία εποπτεία με όλες τις ε, εναλλακτικές λύσεις και για τα ερωτικά προγράμματα που επέμονται. Ποιο είναι εκείνο ο οποίο ελέγχει και διασφαλίζει ότι όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον, το public domain, δρούμε σωστά. Ασχολούμαστε με τα φιλόδοξα και έγκριτα και έντιμα μέσα αλλά υπάρχουν και άλλες επιτυχίες και τα, όσα βιώσαμε τα τελευταία 30 χρόνια όπου πολύ καθυστερημένα ε, λάβαμε υπόψη. Για παράδειγμα και σε σχέση με τα βιβλία κάθε δημοσίευμα θα πρέπει να ε, παρέχεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε αντίτυπο, στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη ενώ είναι πολύ σημαντικό για παράδειγμα να δούμε για τα οπτικοακουστικά ότι απουσιάζει πλήρως εδώ η πτυχή των ιδιωτικών καναλιών. Τώρα, το να μην ε, ε, υπάρξει καμία τέτοια δράση μία εβδομάδα ετήσια υπάρχει παρακολούθηση ή ε, μαγνητοσκόπηση. Για παράδειγμα, αν είχαμε π.χ. Ε, στη δεκαετία του 60 τέτοια γεγονότα και είχαμε τέτοιου είδους ε, διαφημίσεις απευθύνω έκκληση για την ελαστικότητα που για το παρελθόν με καθυστέρηση αναπτύξαμε τώρα τουλάχιστον για το παρόν και για το μέλλον να προσέξουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αν ε, αγωνιζόμαστε για να βρούμε την τέλεια διατύπωση Φυσικά σε σχέση με ένα μεγάλο τέτοιο κατάλογο ειδήσεων, εκπομπών, σε σχέση με την εικόνα, μια τεράστια ας το πω έτσι συνιστόσα για το πρόγραμμα στα, στα Euromedia στα, μέσα της δεκαετίας του 90 και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια τέτοια σιζοφρενική τάση όσον αφορά για παράδειγμα τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύξαμε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, η εικόνα να μπορεί να δίνει την ε, πραγματικότητα σε σχέση με τους ε, ε, ηλεκτρονικούς εγκεφάλους. Και είχαμε τη δυνατότητα ψηφιοποίησης σε μεγάλη κλίμακα και δημοσιοποίησης. Χρειαζόμαστε και τα δύο λοιπόν. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστότερη προσέγγιση για την νομική ρύθμιση, ώστε με εικόνες να βλέπουμε ποιο είναι το περιεχόμενο. Και η πλήρης χρήση πρέπει να ακολουθεί, η πλήρης εκμετάλλευση πρέπει νομικά να καθορίζεται ως δυνατότητα ε, συνεισφοράς για τη μόρφωση και την παιδεία. Μέχρι σε αυτά τα πλαίσια μπορεί ένας κατάλογος ή ένα μητρό να μπορεί να λειτουργήσει. Και για τα μικρότερη εμβέλειας προγράμματα, πολλά πράγματα μπόρεσαν να αλλάξουν σε σχέση με την σύγχρονη ιστορία στην Αυστρία επειδή πριν από τον Βαλτχάιμ ε, ως πρόεδρο μπορέσαμε να ασχοληθούμε με αυτή την πτυχή της σύγχρονης ιστορίας και στα αρχεία μας για παράδειγμα τον, τον χρόνο παραγωγής τον μειώσαμε, τον συντμήσαμε για να μπορούμε για παράδειγμα από τα κονδύλια να αντλούμε δυνατότητες να δράσουμε αντί να κάθεται κανείς επί εβδομάδες σε χώρους που δεν έχουν καλό εξοπλισμό για να επιλέξει κανείς ε, το αναγκαίο υλικό. Λοιπόν, μικρής εμβέλειας προγράμματα, μικρής κλίμακας προγράμματα, όπως αυτό το πρόγραμμα ή εγχείρημα για το έτος Verdi Wagner. Να μπορεί κανείς να μαθαίνει, παίζοντας, ε, ενασχολούμενος ε, με τέτοιου είδους, ε, ας το πω θέματα για την παιδεία και την εκπαίδευση. Θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία με τέτοια μικρά προγράμματα αν θέλουμε να συγκρίνουμε αυτή την προσέγγιση με μια ολιστική, σφαιρική προσέγγιση. Και εδώ, ως όπου τα πράγματα και στο YouTube εμείς είμαστε οι πειρατές εκεί όπου με, βλέπουμε ότι εκπέμπονται εκπομπές ε, νοσταλγικού χαρακτήρα εντός εισαγωγικών σε 30 ας το πω έτσι εκπομπές και χωρίς οποιαδήποτε νομική κάλυψη αυτά αναμεταδίδονται μέσω του YouTube. Του YouTube. Αυτό είναι ψηφιακή πειρατεία και πρέπει έτσι να κατανομαστεί και να καταγγελθεί. Δεν μπορεί να γίνεται λοιπόν κάτι τέτοιο. Αλλά όταν έχουμε τέτοιου είδους εικόνες που εκπέμπονται σε τέτοια προγράμματα θα πρέπει να γίνονται προς όφελος του συμφέροντος και να μην αγνοείται η διάσταση του ε, κοινού συμφέροντος public domain εις βάρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, χαίρομαι τώρα που μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Έκερ ακόμα από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οπτικοακουστικά και τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες για την ενημέρωση. Έχουμε μπροστά μας ένα βουνό που πρέπει να ανεβούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει μόνο στους πρόποδες. Λοιπόν, ως προς την ψηφιοποίηση η κατάσταση των πραγμάτων είναι εμβριακή. 10 με 15% έχουμε κάνει, αν και πιστεύω ότι πρόκειται για ακόμα χαμηλότερο ποσοστό. Και τούτο διότι δεν έχουμε συμπεριλάβει τα διάστατα αντικείμενα, αρχαιολογικά αντικείμενα, γλυπτά κλπ. Δεν έχουμε καν, δεν έχουμε καν συνειδητοποιήσει ότι αποτελούν τμήμα τη πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε το βουνό είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι εκτιμούσαμε στην αρχή. Αυτό είναι το πρώτο. Έχω μια σύσταση προς τους βουλευτές, ε, προς τα κρατημέλη με συγχωρείτε, για την ψηφιοποίηση. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, Πρόκειται για 27 διαφορετικές χώρες και μάλιστα ακόμα στην κάθε χώρα, εντός της κάθε χώρας έχουμε διαφορετικούς παίκτες, διαφορετικές καταστάσεις, πρωτοβουλίες κλπ. Ξεκινούμε μια μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας θα τεθούν κάποια στιγμή για να δούμε πού είμαστε από πλευράς ψηφιοποίησης. Άρα, καταρχήν, η βάση δεδομένων είναι μικρή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει την ψηφιοποίηση. Και εδώ βεβαίω ιδιώτες όπως η Google διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Στη σχετική οδηγία έχουμε προσθέσει διάταξη η οποία αφορά το πώ ακριβώ θα διαχειριστούμε τι σχετικέ συμφωνίε. Χρειάζεται σύμπραξη δημόσιου ιδρύκου τομέα σίγουρα για να προχωρήσουμε. Το ερώτημα είναι σε τι πλαίσιο. Άλλο ένα πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά. Η Ευρωπαϊκή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ψηφιοποιεί. Κάνει πολλή δουλειά η Ευρωπαϊκή η οποία προκαλεί, οδηγεί σε ψηφιοποίηση και υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά η Ευρωπαϊκή αξιοποιεί έργα που ανήκουν σε πολιτιστικούς οργανισμούς. Η όμως δεν κατέχει ψηφιακά αντικείμενα ίδια. Κατέχει μεταδεδομένα, τα οποία αναφέρονται ακριβώς σε ψηφιοποιημένα πολιτιστικά αντικείμενα. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στα 22 εκατομμύρια, όντως που ανήκουν στη δημόσια σφαίρα. Η Ευρωπαϊκή κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Ομαδοποιεί το περιεχόμενο, Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιο να ψάξει στο συγκεκριμένο μουσείο, στη συγκεκριμένη χώρα. Όχι. Η Ευρωπαίνα θα σα πάει σε όλα τα συγκεκριμένα αντικείμενα σε όλη την Ευρώπη. Είτε είναι σε ένα Βρετανικό μουσείο, είτε σε ένα Βαλγικό μουσείο, είτε σε ένα Πορτογαλικό μουσείο. Αυτό κάνει η Ευρωπαίνα και αυτό είναι η πολύτιμη συμβολή τη. Η Ευρωπαίνα επίση προάγει την τυποποίηση. και αυτό ακολουθώντας πρωτοβουλία αμερικανική. Ό,τι ψηφιποιείται τώρα βεβαίως μπορεί να γίνει διαθέσιμο Η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου είναι ένα δεν λύνει το πρόβλημα φυσικά και έχουμε και άλλη μια πρόταση στο τραπέζι που είναι η διαφάνεια, η οδηγία για τη διαφάνεια για, τη, για τους οργανισμούς συλλογικών δικαιωμάτων. Και πάλι όμως δεν λύνουμε το πρόβλημα που έχουν προκειμένου. Αν δούμε τώρα την κληρονομιά των ταινιών, μόνο 1,5% αυτών έχουν ψηφιοποιηθεί. Μόνο 1,5%. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών είναι διαθέσιμα διαδικτυακά. Τα μη διαθέσιμα και τα μη ψηφιοποιημένα είναι εκτός εμπορίου, δηλαδή προστατεύονται, αλλά εν γέννη δεν χρησιμοποιούνται καν. Αυτή λοιπόν η περιουσία που βρίσκεται εκτός εμπορίου πρέπει κάπως να μπει στο κύκλωμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι και για αυτήν την περιουσία, για αυτά τα στοιχεία, ε, εξυγχρονίζοντας το σύστημα προστασίας. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να πάμε από τους πρόποδες στην κορυφή του βουνού. Η οδηγία PSI πρέπει να εγκριθεί καταρχήν. Πρέπει να θεσπίσουμε μια σύσταση για την αρχαιοποίηση, ψηφιοποίηση και το καθεξής. Αυτά για το 2013. Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή να γίνει πιο ελκυστική. Και ένα άλλο κρίσιμο βήμα είναι η χρηματοδότηση στα πλαίσια του επομένου πολιτού χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020. Η Ευρωπαϊκή θα χρηματοδοτηθεί μέσω του μηχανισμού Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη και χαίρομαι διότι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας διατηρείται η χρηματοδότηση για τον σχετικό μηχανισμό, άρα παίρνουμε πλέον στην τελική φάση της σχετικής συζήτησης. Και έτσι θα εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την Ευρωπαϊκή και άλλες υπηρεσίες στο μέλλον. Τέλος, εξίσου σημαντικό, πρέπει το 2013 να συνεργαστούμε με την βιομηχανία, με τον ιδιωτικό τομέα για να θεσπίσουμε ένα μοντέλο χωρίς αδειών, πιο προοδευτικό, πιο ευέλικτο, ανεξαρτήτως της αναθεώρησης της προστασίας των δικαιωμάτων, κάτι πάνω στο οποίο δουλεύει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κυπριακή Προεδρία εκπροσωπείται από τον κύριο Σολομού. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο να παρέμβετε. thanks, Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Πρόεδρε, για τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, Πολιτισμού, αγαπητοί συνάδελφοι, Κυπριακή Προεδρία θέλει να ευχαριστήσει για την πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για τις προς ευκαιρίες ε, για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Κυπριακή Προεδρία ομόθυμα και ομόφωνα θεωρεί ότι αυτές οι ευκαιρίες ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πολιτιστική κληρονομιά. Θεωρούμε ότι έχει τρεις διαστάσεις αυτό το ζήτημα. Τη νομική διάσταση, τις υποδομές και την χρηματοδότηση ως άξονες και μια σφαιρικότερη διάσταση που συνδέεται με τις δομές όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα που θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την κοινωνία της πληροφορίας θα ήθελα να τονίσω σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν για το, τις μελλοντικές εξελίξεις και από πλευράς του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα για την επισκόπηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου όσον αφορά τον τομέα του, των πολιτιστικών θεμάτων και της διασφάλισης ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το τελευταίο Συμβούλιο που έγινε Δεύτερον, θα ήθελα επίσης κάποιες δράσεις να αναφέρω από το τρέχον που συνδέονται με την πρόταση στην οποία έχουμε καταλήξει για την Connecting Europe Facility, την, το μέσο διασύνδεσης ε, για την Ευρώπη και την πρόσβαση στην πολιτισμική πολυμορφία. Με πρίσμα αυτή την πολιτισμική ε, πολυμορφία πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις ε, προηγούμενες αλλά και τις σημερινές έπτυχες και δράσεις λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές αυτές προοπτικές. Εν τέλει θέλω να, να αναφερθώ σε μια πιο μακροπρόθεσμη ε, συνιστόσα για τον, την ψηφιακή εποχή που απασχολεί το Συμβούλιο που όμως δυστυχώς ε, δεν εγκρίθηκε και κατά τη διάρκεια αυτής της δικής μας Προεδρίας μέχρι σήμερα. Τα συμπεράσματα λοιπόν του Συμβουλίου για την ψηφιοποίηση και για την, τα πολιτιστικά στοιχεία από πλευρά ε, του Συμβουλίου του Μαΐου ανανεώνουν τις τα προηγούμενα συμπεράσματα του Νοεμβρίου 2006 ε, καθώς επίσης ε, και στοιχεία τα οποία εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη μελλοντικών δράσεων για την Ευρωπαϊκή σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2010 ευχαριστώ. και κατά άλλα, αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θέλουν να ανανεώσουν την προαγωγή προς μια επιτυχή ψηφιοποίηση όσον αφορά τις διεργασίες, καθώς επίσης και ένα ε, πρόγραμμα σε σχέση με τις συστάσεις ε, που υπευλήθησαν τον Οκτώβριο του 2011. Αυτές οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 εμπεριέχουν επικαιροποιημένα μέτρα και δράσεις για την ψηφιοποίηση και την διάθεση στο διαδίκτυο πολιτιστικών στοιχείων και υλικού γενικότερα όσον αφορά και την πολυμορφοποίηση που αποτελεί όρο εκ των όνου κάνεφε για την δυνατότητα να υπάρχει διάθεση και διάχυση αυτού του υλικού. Επίσης ε, η ψηφιοποίηση και η διασφάλιση μέσω ψηφιοποίησης δημιουργούν ε, αξιόλογα στοιχεία από πλευράς ε, του πολιτισμικού υλικού. Το να γίνουν αυτά τα στοιχεία πολύτιμα στοιχεία μέσα σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεισφέρουμε έτσι μέσα σε ένα πλαίσιο καινοτομία στις δράσεις μας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας τομέας που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα άξονα αηφορίας, αηφορία στην ανάπτυξη, βιωσιμότητα στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα όσον αφορά το παράτημα σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ε, περιέχει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα με προτεραιότητες από των κρατών μελών για δράσεις κατά τα επόμενα τρία έτη από τα κράτη-μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη ε, τις προκλήσεις ε, δημοσιονομικά και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των θεμάτων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να δούμε τις ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσπελασιμότητας και διάθεσης αυτού του πολιτιστικού υλικού στο κοινό και της περαιτέρω επεξεργασίας και ολοκλήρωσης της πρωτοβουλίας Ευρωπαίανα η χρηματοδότηση από πλευράς ε, της ε, ΕΕ για την διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο τέτοιου είδους ε, στοιχείων μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής όπως, μόλις, όπως αναφέρθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί τμήμα της πρωτοβουλίας του μέσου διασύνδεσης της Ευρώπης, Connecting Europe Facility. Πράγματι, αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν τμήμα ε, των υποδομών του κεφαλαίου υποδομών για την ψηφιοποίηση από πλευρά ε, των δράσεών μας για το μέσο της ε, διασύνδεσης της Ευρώπης λαμβάνοντας υπόψη και τον τομέα για παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών και των κονδυλίων έχει εγγράψει ενδεικτικά ποσά η Κυπριακή Προεδρία για αυτές τις δράσεις, ώστε να υπάρξει μια δυνατότητα να διαμορφωθεί ένας προϋπολογισμός όσον αφορά τα α, ε, τηλεπικοινωνιακά και να μην υπάρξει σημαντική περικοπή όσον αφορά τις ε, προτάσεις ε, Αυτά είναι όμως ενδεικτικά ποσά τα οποία εναπόκεινται στην διαπραγμάτευση για να επιβεβαιωθούν. Το τελικό ποσό το οποίο θα διατεθεί σε σχέση με τις χρήσεις τηλεπικοινωνιακές χρήσεις θα πρέπει να αναμείνουμε να διαμορφωθεί. Και σε σχέση με το μέρος αυτό το οποίο τμήμα του Connecting Europe Facility που έχει τη σπουδαιότητά του για τα θέματα τα οποία συζητούμε σήμερα είναι με στόχο να συνεχιστούν οι συζητήσεις μέχρι ότου να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις επί της ε, πρικοδότησης των κονδυλίων. Για να δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα για την Ευρώπη, που αποτελεί την άλλη πρόταση που απορρέει από την δημόσια ακρόαση, σε πρώτη ανάγνωση, με παρόμοιους ε, συναφείς στόχους που είναι να μπορέσουμε να διευκολύνουμε να υπάρξει πλήρες όφελος από τα θέματα τα πολιτιστικά. Κάποιες εβδομάδες ε, είχαμε συζητήσεις με αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για αυτό το θέμα κατά το παρελθόν. Σύντομα θα ήθελα να αναφέρω κάποια πληροφοριακά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Πράγματι μόνο ενδεικτικά διακόπτεται από την Πρόεδρο. Δεν νομίζω ότι έχουμε τώρα το χρόνο για να ακούσουμε προβληματισμούς για τον προϋπολογισμό από πλευρά σας. Θα ήμουν ευγνώμων. Δεν είναι το ενδιαφέρον για τους επαΐοντες, για τους πραγματογνώμονες το θέμα των κονδυλίων και του προϋπολογισμού. Θα το συζητήσουμε σε άλλη συνάντηση. Ολοκληρώσατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ολοκλήρωσα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνεδρίασης. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους πραγματογνώμονες. Μας άνοιξαν τα μάτια περισσότερο για να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για το εύρος των θεμάτων που... Παρακαλώ, μπορείτε να συζητήσετε, να σβήσετε το μικρόφωνο από την Κυπριακή Προεδρία γιατί Μάλιστα, ευχαριστώ. Μπορώ να συνεχίσω στα γερμανικά. Ευχαριστώ λοιπόν στους πραγματογνώμονες. Ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητική η συμμετοχή και παρέμβασή τους. Συνεισφέρατε με ένα πολύ σημαντικό τρόπο και θετικά στις συζητήσεις μας και στο, στους προβληματισμούς μας. Έχουμε προκλήσεις ενώπιον μας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτές τις προκλήσεις φωτίσατε και φωτίστηκαν όσον αφορά τα μητρώα και αρχεία ε, ψηφιοποίησης ε, στο διαδίκτυο online. Ακούσαμε για το τι έγινε στο παρελθόν, το data licensing και το copyright και φυσικά νομικές πτυχές και τις διάφορες μεθόδους. Πώς, διαφορά, πώς διαφορετικά μπορεί η πολιτιστική κληρονομιά μέσω αυτών των links ε, να προστατευτεί. Έχουμε ένα ολόκληρο βουνό, υψηλό, ψηλό βουνό μπροστά μας που πρέπει να ξεπεράσουμε, να διαβούμε. Όμως υπάρχει μια βραδύτητα που ας το πω έτσι όταν προσπαθούμε να αναρριχηθούμε, να ανέβουμε σε αυτό το βουνό, μας ξεπερνούν πάλι τα γεγονότα. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κρατικό μόρφωμα. Αποτελείται, συναπαρτίζεται από 27 κράτη-μέλη και το πρόβλημα είναι ότι από τα λάθη μας θα έπρεπε να μαθαίναμε. Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Συζητάμε για αυτά τα λάθη και ξέρουμε ότι πρέπει να μάθουμε από αυτά, αλλά τα μέσα και ο ρυθμός τους είναι βραδύτατος και βραδύτατα. Και αν αυτά δεν υλοποιούνται και δεν υλοποιούνται και από τα κράτη είναι και αυτό είναι επιπρόσθετο πρόβλημα. Και αν στοχεύουμε στο 2014 για μια συγκεκριμένη οδηγία, μέχρι να εφαρμοστεί θα περάσουν και άλλα περισσότερα χρόνια. Με άλλα λόγια, πρέπει ουσιαστικά αυτούς που μας παρακολύουν, δηλαδή τις εθνικές κυβερνήσεις, που δεν έχουν προχωρήσει ώστε να έχουν μάθει από τα σφάλμα τους, να έχουν συναγάγει τα συμπεράσματα τα σφάλματά τους, όπως εσείς ρητά αναφέρατε σήμερα, πρέπει να ασκήσουμε επιρροή και πίεση στους εθνικούς πολιτικούς εκπροσώπους και τις κυβερνήσεις, ώστε ταχύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσουν, ώστε να διευθετηθούν ταχύτερα τα πράγματα τα οποία εκκρεμούν. Διότι διαφορετικά, όπως ακούσαμε, για την Ευρωπαϊκή και την πρόοδο που έχει επιτελεστεί. Πολλές φορές κάποια αστεία γίνονται. Τι λένε, έχετε την Ευρωπαϊάνα, τι γίνεται με αυτήν. Λοιπόν, για τα όσα αναφέρθηκαν ότι υπάρχει ένα πρότυπο το οποίο αντιγράφουν οι Αμερικανοί. Πρέπει αυτό το πρότυπο να το κάνουμε πιο θελκτικό, πιο ελκυστικό. Πρέπει να βοηθήσουμε, να γίνει κάτι αποτελεσματικό και να βοηθήσουμε για αυτούς τους καταλόγους ή μητρώα. Εγώ θα έλεγα, θα τα αποκαλούσα καταλόγους. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στους καταλόγους, στα μητρώα αυτά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν κάτι κάποιο θέλει από αυτούς τους καταλόγους, έστω να πληρώνει κάποιο αντίτιμο. Αλλά είναι απλά πράγματα. Είμαι πρακτικός άνθρωπος. Δεν είμαι νομομαθής, ε, ούτε θέλω να περιπλακούν τα πράγματα. Ανατριχιάζω όταν βλέπω πόσο νομικίστικα ρυθμίζονται κάποια πράγματα που περιπλέκουν ανούσια την ουσία. Εξαιρετικά μας τα υπεξηγήσατε και σας ευχαριστούμε. Και ζητώ συγγνώμη για τους συναδέλφους που απουσιάζουν, δεν είναι τεμπέληδες και δεν αδιαφορούν, αλλά πραγματικά βρίσκονται σε κοινοβουλευτικές επιτροπές που έπρεπε να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν σε ψηφοφορίες, γι' αυτό απουσιάζουν. Να επισημάνω κάτι το briefing αυτό είναι μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό γεγονός. Έγινε πολλή δουλειά για την πρόσβαση καταναλωτών ε, online και την προσπελασιμότητα του πολιτισμικού και πολιτιστικού υλικού στην ψηφιοποίηση στο διαδίκτυο. Εξαιρετική δουλειά είναι αυτή θα έπρεπε να το δείτε και να το λάβετε υπόψη ως επαΐοντες επ' αυτού. Ίσως θα διευκολύνει τη δουλειά για μας και για σας. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι συνάδελφοι είναι ελεύθεροι τώρα, εκτός από εκείνους που θα συμμετάχουν στη συνάντηση των συντονιστών. Και έληξε η συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat> Θα ξανασυναντηθούμε. Θα πρόκειται για θέματα εκπαίδευσης. Yes Europe, όχι για το, Erasmus, ε, το έρασμο για όλους, αλλά για το Yes Europe. Αν έτσι λοιπόν ε, προσπαθήσετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα με αυτές ε, τις εικόνες που είναι καλές, σας ευχαριστώ. Έχετε όλοι αυτά τα φύλλα, αυτά τα χαρτιά.